Okay, colleagues, if I can start. Αγαπητοί συνάδελφοι, βέβαια δεν είναι πολύ εδώ, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Επειδή τελειώνει η θητεία μου Προέδρου, δεν θέλω να πακτήσω κακές συνήθειες. Έχετε το σχέδιο τη διάταξης. Συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έγκριση των πρακτικών 22-23 Τετάρτου 6-7 Μαΐου. Εντάξει. Ωραία. Πριν περάσουμε στην έκθεση του Ντομινίκ, ένας από μάλλον μία από τις βοηθούς, ε, η Τζούντιθ που έχει ε, δουλέψει πάρα πολύ καιρό και επιστρέφει στην Αυστρία για να γίνει δικαστήνα. Ελπίζω λοιπόν ότι η θητεία της εδώ τη βοήθησε, αλλά μήπως θα πεις κάτι, Ιωάν. Ευχαριστώ που αναφέρατε αυτό το λυπηρό γεγονός Ε, η Τζούντιτ με βοήθησε πολύ. Τώρα που φεύγει δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί η δουλειά μου. Αλλά θα ήθελα να πω ευχαριστώ πολύ στη Τζούντιτ για τη θαυμάσια εργασία και για τη φιλία σου. Ε, όντως ήταν θαυμάσια συνεργασία μας και η εμπειρία της συνεργασίας μας. Τζούντιθ, ε, σου ευχόμαστε όλοι τα καλύτερα στη νέα σου σταδιοδρομία. Αν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην Αυστρία, έχουμε επαφή. Εάν αν δεις έναν ε, ε, ηλικιωμένο ευρωβουλευτή μπροστά σου στην Αυστρία, ελπίζω να με θυμηθείς. Επόμενο θέμα, η έκθεση Ντομινίκ Ρίκε, η οδηγία για τον εξοπλισμό των ε, πλοίων, εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Παρακαλώ, Ντομινίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων. Όχι βέβαια η έκθεση αυτή δεν ε, δεν εξετάζει τα πάντα, αλλά κοιτάζει κυρίως ε, τα βοηθήματα ναυσιπλοείας, τα μέσα πυρόσβεσης, όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί, οι διεθνείς κανονισμοί απαιτούν ε, τα κράτη να ελέγχουν τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας αυτών των εξοπλισμών. Υπάρχει λοιπόν μια οδηγία η οποία επέτρεψε να μειωθούν οι σοβαρές ε, διαφορές που υπήρχαν από κράτος σε κράτος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμη προβλήματα. Καθυστερεί τη μεταγραφή της νομοθεσίας, αλλά και οι εθνικοί οργανισμοί που ελέγχουν ε, κατά πόσον ε, συμμορφούνται οι εξοπλισμοί αυτοί λειτουργούν με άνισο τρόπο και υπάρχουν και διάφορα κενά στην αγορά. Αυτές οι διαφορές σημαίνει ότι υπήρχαν και διαφορές στην ασφάλεια στα πλοία. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν είναι σκόπιμη <clears throat> για να καλύψει ένα κενό, να επιτρέψει να ενισχύσουμε την νομική διαφάνεια και για τις επιχειρήσεις που ε, κατασκευάζουν και πουλούν αυτό το εξοπλισμό, αλλά και την ασφάλεια ε, εμπλών. Καλή λοιπόν αυτή η οδηγία. Θα προτείνω μια σειρά από τροπολογίες που στοχεύουν να διευκρινίσουν κάποιες ασάφειες όσον αφορά τη διάρκεια για την οποία πρέπει, ε, διάρκεια κατά την οποία πρέπει να τηρούνται κάποια έγγραφα και άλλα τεχνικά στοιχεία. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει αυτό το σήμα του πιδαλίου. Δεν είναι το ίδιο το πιδάλιο, είναι ένα σήμα που έχει ένα πιδάλιο επάνω που έχει να κάνει με το κατά πόσον ε, συμμορφούνται με τις, ε, με τις προδιαγραφές για να ελέγχουμε εάν ε, υπάρχουν απομιμήσεις διότι και στον τομέα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα οι απομιμήσεις θέλουμε να δούμε πότε θα αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό το παλιό ε, σχήμα. Επίσης ε, ο έλεγχος της αγοράς πρέπει να είναι ανάλογος ε, με το περιεχόμενο του ελέγχου, ιδιαίτερα η δειγματοληψία που ζητούν τα κράτη. Γιατί αν είναι υπερβολική αυτή η έλεγχη μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις κόστους. Και φυσικά ε, για τα υπόλοιπα θα έχω την ε, συνήθη στάση όσον αφορά τις κατοικουσιοδότης πράξης του Κοινοβουλίου. Αυτά για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν από πλευρά σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία του. Συνολικά Συμφωνούμε και με την πρόταση της Επιτροπής και με αυτά που έγραψε ο κύριος Ρικέ. Δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν τρία σημεία που θέλω να σχολιάσω. Για τα δύο ακόμη είμαστε σε φάση επεξεργασίας και το τρίτο οπωσδήποτε θα υποβάλουμε τροπολογία. Πρώτον, ο έλεγχος ε, ε της συμμόρφωσης από τις ε, πιστοποιημένες αρχές. Αυτές οι αρχές πρέπει να διαπιστώνουν ότι ο εξοπλισμός των πλοίων συμμορφώνεται με τις οδηγίες και όλα τα άλλα ε, ισχύοντα διεθνή μέσα και προδιαγραφές. Είναι τεχνικά όλα αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρμοδιότητα να κρίνουμε κατά πόσον ισχύουν οι προδιαγραφές και τα διπλώματα τεχνίας, τα πρότυπα, θα πρέπει να δούμε εάν έχει έννοια εδώ να ενισχύσουμε την, ε, τον έλεγχό μας. Δεύτερον, η παροχή πληροφοριών προς αυτές τις αρχές δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι αυτές οι εξοδοτημένες αρχές ενημερώνουν τις περαιτέρω αρχές για το εάν όλα βαίνουν καλώς. Αυτή η πληροφόρηση για τα θετικά και αρνητικά των ελέγχων πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται. Για να ελέγξουμε ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό, εάν αυτός ο έλεγχος γίνει μόνο από έναν οργανισμό, Υπάρχει πρόβλημα εάν και κατά πόσον είναι ο καλύτερος αυτός ο έλεγχος, εάν ε, προσφέρει την αναγκαία προστιθέμενη αξία. Πρέπει να το εξετάσουμε. Το τρίτο σημείο, τουλάχιστον για μένα όμως, είναι σαφές. Η πρόταση καθορίζει ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να διατηρούν ένα αντίγραφο για 10 χρόνια του εντύπου που πιστοποιεί, να, πιστοποιεί την συμμόρφωση και επίσης ε, και τα σκάφη. Τα πλοία πρέπει να τηρούν ένα τέτοιο αντίγραφο. Πρέπει λοιπόν και ο παραγωγός και η αρχή να έχει αυτό το αντίγραφο. Νομίζω ότι κάνουμε δύο φορές την ίδια δουλειά, δεν χρειάζεται να διατηρήσουμε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με την άποψη του κυρίου Ρικέ και ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, από πλευρά ε, ε, φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ για την εργασία του καταρχάς. Δεν θα σας ε, εκπλήξει ότι και ο κύριος Φλέκενστάιν και εγώ είμαστε από τη Βόρεια Γερμανία, άρα μιλήσαμε με τους ίδιους συνομιλητές. Πρέπει να δούμε τι έχει έννοια για να βελτιωθεί η ασφάλεια των πλοίων και να μπορούν να αντιδρούν καλύτερα σε ατυχήματα που είναι σκόπιμο να υπάρχουν γραφειοκρατικές απαιτήσεις και που δεν είναι σκόπιμο. Έχω ακριβώς ε, τα ίδια θέματα να τονίσω με τον κύριο Φλέκενστάιν. Αυτό το θέμα για τα έντυπα και τι ελέγχους πρέπει να κάνουν οι εξοδοτημένες αρχές ε, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτές οι αρχές να κάνουν τον ε, αστυνομικό έλεγχο των προτύπων και προδιαγραφών το εξετάζουμε το θέμα αυτό και κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλουμε τροπολογία για τα αντίγραφα, το ότι πρέπει να τηρούν, τηρούνται αντίγραφα σε δύο διαφορετικά σημεία. Νομίζω ότι ως Ευρώπη θέλουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να ισχύει και για τον εξοπλισμό των πλοίων και κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω. Δηλαδή, στο άρθρο 13.1 αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι εξισοδοτημένοι ε, αν ε, κάποιος εξοπλισμός και να χορηγούνται κάποιες εξοδοτήσεις ε, αν κάποια, κάποιοι εξοπλισμοί παράγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό τους ούτως ή άλλως ήδη παράγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν ε, δυνατό να υπάρχουν αυτές οι εξοδοτήσεις για όλα αυτά τα προϊόντα. Πρέπει να ε, αναρωτηθούμε αν αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βελτιωθούν προδιαγραφές ελέγχου πολλές φορές δεν είναι αρκετά δεσμευτικές. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπάρχουν εξαιρέσεις και ε, θα πρέπει να γίνει ταχύτερα η μεταγραφή στο εθνικό δίκαιο. Ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραχάραξης ε, των πιστοποιητικών. Πρέπει να ισχύουν παγκοσμίω όλα αυτά. Ε, κατά βάση όμως συμφωνούμε με τον εισηγητή τον ε, συγχαίρω για τη θαυμάσια εργασία του, στην οποία και εμεί συμβάλαμε και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Μπράτφορντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω να κάνω δυο-τρει παρατηρήσει που είναι τεχνικού χαρακτήρα κυρίω. Καταρχά ένα, για τα οποία ένα σημείο για το οποίο έχω μεγάλη επιφύλαξη σε σχέση με αυτή την πρόταση είναι σαν να υφέρπει μια επέκταση των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν και αυτό φαίνεται όταν δούμε την πρόταση για τις κατεξουσιοδότηση πράξης και όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο και όσον αφορά τον τρόπο που υποβάλλονται και ε, θα ήθελα αυτού του είδους στην αρχή, αν θέλετε, να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Επίσης, για κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα, είναι ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα σε σχέση με αυτό το οποίο ήδη υπάρχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Θάλασσας. Χρειαζόμαστε παγκόσμια πρότυπα εδώ και αυτό το οποίο δεν θέλω να συμβεί είναι είτε να έρθουμε σε αντίθεση είτε να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα ε, σε σχέση με αυτό το οποίο ήδη υπάρχει. Αυτές είναι οι βασικές ανησυχίες όπως επίσης και το θέμα του κόστους. Πουθενά στα έγγραφα τα οποία έχω δει εγώ τουλάχιστον δεν αναφέρεται ε, κάποιος υπολογισμός του κόστους όπως χάρη για την αντικατάσταση του του πιδαλιοσχήμου σήματος. Όλα αυτά, εάν τα λάβουμε υπόψη μας και παράλληλα και με τις άλλες προτάσεις που γίνονται εδώ, κοστίζουν τεράστια ποσά. Επομένως έχω κάποιες επιφυλάξεις και ελπίζω ότι όλα αυτά ο κύριος Ρικέ θα τα λάβει υπόψη του όταν ε, λάβει υπόψη και τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν στην ε, αίθουσα αυτή. Ευχαριστώ κύριο Κέρν Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον Ντομινίκ Ρικέ και τους Κιώδης για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Φυσικά όλα τα κράτη που έχουν ναυτιλία εκπροσωπούνται στα διεθνή όργανα και τον IMO, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, Οπωσδήποτε ε, λοιπόν συμμορφούνται με τον κανονισμό για την ασφάλεια εν πλώ, όπου υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές, ποια σωστικά μέσα πρέπει να έχουν τα πλοία, για τα, εμπορικά, τα εμπορικά πλοία, τα φορτηγά πλοία, τα επιβατικά πλοία, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου οι προδιαγραφές, όπως είπε και ο κ. Φλέκενστάιν, που απαιτούνται οι προδιαγραφές λοιπόν αυτές, δεν ελέγχονται και άρα δεν τηρούνται όσον αφορά τα σωστικά μέσα, τα βοηθήματα της ναυσιπλοείας, τους ε, μηχανισμούς για την σταθερότητα των ε, σκαφών. Δεν ελέγχεται αν υπάρχουν τα αναγκαία πιστοποιητικά και εάν τηρούνται οι προδιαγραφές. Και ποιο είναι το περιεχόμενο των προτύπων αυτών. Γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί, αυτοί οι εξοπλισμοί για όλα αυτά, τα φορτηγά, τα επιβατικά, τα πλοία κρουαζιέρας, τα ferry boat, εάν τηρούνται όλα αυτά τα οχηματαγωγά. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ισχύουν όλα αυτά γιατί ορισμένοι μηχανισμοί που ε, παράγονται σε τρίτες χώρες δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επιβατών, των πληρωμάτων και να αποφύγουμε τα ε, μεγάλης διάστασης ε, ατυχήματα εμπλό, συγκρούσεις. Φυσικά δεν θέλουμε να υπάρξει υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά πρέπει να γίνουν αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Καραμίτσος, εξ ονόματος της Κομισιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ για την εξαιρετική του έκθεση, η οποία είναι ισορροπημένη, είναι λογική και οι περισσότερες των τροπολογιών μπορεί να γίνουν δεκτές. Για να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία, και αυτό για δύο λόγους, ο ένας είναι η απλούστευση, πιστεύω ότι η πρόταση αυτό το οποίο θέλει είναι να δημιουργήσει ένα απλό σύστημα έτσι ώστε να, μετατεθούν, να μπορούν να μεταφερθούν οι διατάξεις σχετικές με την ε, παγκόσμια ναυτιλία στην ε, ε, κοινοτική νομοθεσία και στην νομοθεσία των κρατών μελών και αυτό Θέλουμε να δημιουργήσουμε επίσης και ένα κάποιο πλεονέκτημα ε, για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, Ευρωπαίους ναυπηγούς, διότι υπάρχει πάρα πολύ εξοπλισμός ο οποίος κυκλοφορεί και ο οποίος δεν είναι σωστός, δεν, είναι, δεν παρουσιάζεται με τον σωστό τρόπο. Έτσι, ε, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι οτιδήποτε μπαίνει πάνω στα πλοία να είναι ο κατάλληλος εξοπλισμός. Η οδηγία ε, δημιουργεί μια κάποια σειρά αλλαγών που συμβαδίζουν με την συνθήκη της Λισαβόνας και επιταχύνει επίσης και τον σεβασμό των παγκοσμίων προτύπων όταν τεθεί σε εφαρμογή και απλουστεύει επίσης και την ε, ε, όλη κατάσταση και για τους Ευρωπαίους ναυπηγούς και τα κράτη-μέλη. Ε, η Ιρλανδική Προεδρία βέβαια πρέπει να έχει κάνει μάλλον τεράστια πρόοδο πριν από το Συμβούλιο το οποίο θα, των Υπουργών το οποίο θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία επί των θεμάτων αρχής θα επιτευχθεί γρήγορα, όπως ε, όμως ένας από τους ομιλητές έθιξε ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τις κατεξιοδότηση πράξεις και για την ε, θεσμική τους αξία αν θέλετε. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τα μάτια ανοιχτά, να δούμε τι μπορεί να γίνει, μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα εδώ. Αυτά είναι τα βασικά. Ε, πιστεύω ότι η έκθεση είναι καλά, ισορροπημένη και μπορούμε να πετύχουμε ε, πρόοδο σε σύντομο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καραμίτσο. Ντομινίκ, θέλεις να προσθέσεις ε, κάτι? Όχι, Πρόεδρε, σημείωσα προσεκτικά το σύνολο των παρατηρήσεων. Θα το συζητήσουμε και με τους σκιώδεις εισηγητές ε, σύντομα, επομένως θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τις, την ε, υποβολή τροπολογιών είναι το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου και 9 Ιουλίου προτιθέμενα να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και θα περάσει από την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου 2013. Επομένως, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 5 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Ο κύριος Κουσιέρη έχει το λόγο ως συντάκτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή την οποία ζήτησε η Επιτροπή αφορά ε, αφορά το σημείο αυτό για τις επιπτώσεις. Ε, εμείς θα συντάξουμε την γνωμοδότηση μεν, επί της ουσίας όμως υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Λοιπόν, ε, εδώ τροποποιείται η οδηγία 2011 του 92 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ε, για ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Εδώ υπάρχουν κάποιες νομικές ε, επιπτώσεις και κάποιες νομικές δεσμεύσεις ε, για, για, τα, γιατί τα έργα αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές, ε, να επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον. Τέλος πάντων, η οδηγία δεν είναι αμφιλεγόμενη και από τον καιρό που υιοθετήθηκε πριν από 25 χρόνια ε, αυξήθηκε και ο αριθμός των προβλημάτων, των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ε, πρέπει να εξεταστούν, αλλά και ο αριθμός των έργων. Ε, η οδηγία αυτή προσαρμόστηκε και τροποποιήθηκε πολλές φορές, όμως δεν, ε, ποτέ δεν έλαβε υπόψη όλες αυτές τις ριζικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα έκτοτε. Γι' αυτό η Κομισιό θέλει να προσαρμόσει την οδηγία αυτή σε αυτό το νέο πολιτικό, οικονομικό και τεχνικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τις τροπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί και με το όλο πλαίσιο γενικότερα το οποίο δημιουργείται πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε τα κενά τα οποία έχει η διαδικασία, τον έλεγχο, την ποιότητα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και τον κίνδυνο να υπάρχουν κάποιες συμβατότητες. Όσον αφορά την ε, επιτροπή, τα θέματα που αφορούν την Επιτροπή ε, Μεταφορών, ε, πιστεύω ότι οι προτάσεις που υποβάλλει η Κομισιό είναι σωστές, λόγω ακριβώς και του διασυνοριακού χαρακτήρα που έχουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η αλλαγή του, του κλίματος και ο κίνδυνος καταστροφών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει ε, να υπάρξει αυτή η ευθυγράμμιση όλων των προτύπων και των ε, ε, διατάξεων, των νομοθετικών διατάξεων, διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνει και η ασφάλεια στην Ευρώπη. Προτείνω επομένως μια σειρά βέβαια τροπολογιών όπου θα λαμβάνει υπόψη αυτές, τις, αυτές μου τις προσδοκίες αν θέλετε ή τις απαιτήσει. Ε, αυτό το οποίο θέλω είναι να αναγνωρίσουμε ακριβώς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν αυτά τα διασυνοριακά project, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για τις μεταφορές ε, στην Ευρώπη. Η αρχική οδηγία λάμβανε υπόψη τα project αυτά, τα οποία έχουν διασυνοριακές ε, επιπτώσεις και σαν ε, συνέπεια πιστεύω ότι είναι σωστό και εμείς να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα δύο συνοριακά έργα. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν αυτά εδώ έτσι ώστε να ε, αυξηθεί αν θέλετε και η, αρμοδιο... και η ευθύνη που έχουν τα κράτη-μέλη να, να... να συντονίσουν τη δράση τους έτσι ώστε να μην δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος. Ε, ένα θέμα το οποίο μας ε, αφορά μένα, αλλά που θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στο κλίμα. Αυτό εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τα θέματα αυτά ανεξάρτητα μεν, όμως οι, οι, μεταφορές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και εδώ. Επίσης εξέτασα και την πτυχή της πρότασης που αφορά τον τουρισμό. Να δούμε και τι επιπτώσεις μπορούμε να έχουμε ε, στον τουρισμό. Υπάρχει η πολιτιστική κληρονομιά των κρατών μελών, ε, υπάρχουν κάποιες ε, τοποθεσίες στα κράτη-μέλη ε, που ζουν από τον τουρισμό και θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε τις περιοχές αυτές να μην υποστούν σοβαρές επιπτώσεις εάν και εφόσον δεν γίνει σωστή η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάποιων έργων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ακούσω τώρα και τι λένε οι συνάδελφοί μου. Ευχαριστώ κύριος Κουμουτσάκος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι βέβαιο ότι η οδηγία ε, ε, που συζητάμε σήμερα παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόστηκε με επιτυχία χρειάζεται ορισμένες προσαρμογές στα νέα δεδομένα διότι τα χρόνια που ίσχυσε διαπιστώθηκαν και αδυναμίες και κενά. Με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτό να οδηγεί τα κράτη-μέλη σε, δικαστική διαδικασία αντιμέτωπο και να προκύπτουν ζητήματα και στο ε, Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επομένως, χρειαζόταν μία προσπάθεια αναθεώρησης και βελτίωσης των ήδη ισχυουσών διατάξεων. Να προσθέσω εδώ και με την ιδιότητα, αν μου επιτρέπετε, του ραπορτέρ στα, ε, για τις κατευθυντήριες αρχές γραμμές των διευρωπαϊκών δικτύων, ότι ο χρόνος στον οποίο ξεκινάει αυτή η συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας περιβαντολογικών επιπτώσεων είναι και πάρα πολύ χρήσιμος και σωστός. Είναι ευτυχή συγκυρία που τώρα που βρισκόμαστε στο στάδιο οριστικοποίησης των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συζητάμε τη συγκεκριμένη οδηγία. Εν κατακλείδη, είμαι σύμφωνος, πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση και αυτό θα πρέπει να καταγραφεί και στη δική μας γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις του συντάκτη της δικής μας ε, γνωμοδότησης. Είναι σωστή η προσέγγιση με την οποία αντιμετωπίζει την πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελα μόνο να θέσω ένα σημείο που μου έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό σε σχέση με τις τροπολογίες που προτείνει. Και αυτό αφορά τις τροπολογίες 7 και 10. Στις τροπολογίες αυτές γίνεται αναφορά στην δυνατότητα του, ε, γίνεται αναφορά στον χρόνο που θα πρέπει να κατατίθενται οι αναλύσεις από τις, ε, και εκτιμήσεις περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Δίδεται στην αρχή ένα τρίμηνο και μετά υπάρχει μια πρόβλεψη αν χρειαστεί παράταση ενός άλλου τριμήνου. Ο συνάδελφος συντάκτης γνωμοδότησης εξαιρεί με απόλυτο τρόπο τα ε, έργα κοινού στρατηγικού ενδιαφέροντος που αποτελούν τμήμα του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου από την δυνατότητα επέκτασης αυτής της προθεσμίας. Λέει ότι στην περίπτωση τέτοιων έργων κοινού ενδιαφέροντος και άρα τμήματος των ευρωπαϊκών δικτύων δεν πρέπει να δίδεται η τρίμηνη παράταση. Αντιλαμβάνομαι το σκοπό της τροπολογίας που είναι να πιέσουμε ώστε τα κράτη να προχωρούν γρήγορα στην υλοποίηση των έργων και των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ παρά να προβληματιστώ με το γεγονός ότι κυρίως αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα και, μεγάλα, και μεγάλης κλίμακος. Επομένως κανείς θα έλεγε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο κάποιων παρατάσεων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα μέσον όρο μεταξύ της θέσης του εισηγητή που λέει καθόλου παράταση και της ανάγκης τέτοια έργα, ε, για τέτοια έργα να υπάρχει μια σχετική ευελιξία. Ε, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση εάν χρησιμοποιήσουμε ως τροπολογία την δικαιολογία της τροπολογίας του. Αντί να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο wording που έχει προτείνει, να υιοθετήσουμε αυτό που λέει ως αιτιολόγηση της τροπολογίας. Σε κάθε περίπτωση το σημείο αυτό νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε σε σε μεταγενέστερο χρόνο, διότι όπως σας είπα αναμένεται, ελπίζω, ενδεχομένως και σήμερα, η οριστικοποίηση του κειμένου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και τότε θα πρέπει να δούμε ώστε να είμαστε συμβατοί με αυτό που θα βάλουμε στην γνωμοδότησή μας με ό,τι θα έχει συμφωνηθεί στο κείμενο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Κατά τα λοιπά συμφωνώ και συγχαίρω τον εισηγητή για την ε, δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Mrs. Meissner. Η κυρία Μάσνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, ο οποίος νομίζω έκανε μια εκτεταμένη εργασία. Φαίνεται στη γνωμοδότηση. Ναι, μένει είναι μόνο γνωμοδότηση, αλλά αφορά πολλούς τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Όπως είδαμε και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, αφορά, αφορά τα, τις ε, διαμεθοριακές ε, μεταφορές Αφορά και τον τουρισμό. Όλα αυτά πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Και εγώ είδα αυτό το θέμα των τροπολογιών για τα άρθρα 7 και 10. Καταλαβαίνω. Βεβαίω, καλό είναι να είμαστε ρεαλιστέ. Να πούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία παράταση, αλλά λειτουργεί αυτό στην πράξη. Γιατί δεν βοηθάει αν αυτό το οποίο απαιτούμε ε, είναι στην ουσία ανέφικτο. Καταλαβαίνω τις προθέσεις του εισηγητή, θέλουμε οπωσδήποτε τα τέντη να προχωρήσουν γρήγορα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτόματες μάλιστα. Γιατί ξέρετε ότι για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χρειάζονται διάφορες ε, μελέτες αντικτύπου, όχι μόνο μία. Κατά τα άλλα όμως, ε, πολλά από αυτά που προτείνει ο τα βρίσκω σωστά και ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ. Και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή και για την καλή συνεργασία. Τον ευχαριστώ πολύ. Είπατε πως είναι θαυμάσια συνεργασία. Ε, Βεβαίω για να υπάρξει θαυμάσια συνεργασία για την οποία ευχαριστήσετε τους Κιώδης ε, πρέπει και ο εισηγητή να είναι διαθέσιμος. Βεβαίω είναι σαφές ότι μας αφορά και η δυνατότητα των, ε, ο τομέας των ε, διαμεθοριακών μεταφορών Οπότε ε, πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνε για να μην κάνει ο ένα από μια μεριά των συνόρων ένα πράγμα και ο άλλο από την άλλη μεριά κάτι άλλο. Βεβαίω και η επίπτωση για το κλίμα είναι σημαντικέ και για μα και η επίπτωση στην βιοπικιλότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πριν από 20-30 χρόνια θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει αυξηθεί πολύ η συνειδητότητα, έχουν γίνει οι συμφωνίε ε, και οι συζητήσει παγκοσμίω για το κλίμα λόγω τη κρίση ε, έχει περάσει δεύτερο πλάνο, αλλά να μην το ξεχνάμε. Τρίτο, Βεβαίω οι μελέτε επιπτώσεων, αντικτύπου, δεν θα πρέπει να αυξάνουν ιδιαίτερα το κόστος. Αλλά στην ουσία το κόστος είναι υψηλότερο εάν δεν προσέχουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Άρα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να τηρείται αυστηρός. Γιατί εάν δεν τηρείται κατόπιν διαπιστώνουμε τις ζημίες. Και στην ουσία μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις μελέτες περιβαλλοντικής ε, ε επίπτωσης. Και στον τομέα του τουρισμού βεβαίως ξέρουμε ότι ο τουρισμός μπορεί να καταστρέψει τον τουρισμό. Πρέπει να είναι βιώσιμος ο τουρισμός διότι Αλλιώς μπορεί να υπάρχουν βραχυπρόθεσμα κέρδη, αλλά μακροπρόθεσμα ζημίες. Ξέρετε τώρα ότι σε τεράστια κομμάτια της ακτής της ε, Μεσογείου δεν πάει πια κανείς. Κέρδισαν για 5-10 χρόνια, αλλά κατόπιν ε, λόγω των ζημιών δεν πάει κανείς. Αυτό είναι σωστό που είπε και η Γκεζίνε Μάισνερ. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά για τον τουρισμό. Κάτι άλλο. Συνάντησα έναν ε, βαβαρό βουλευτή πρόσφατα που ήταν δήμαρχος για πολλά χρόνια στο Στρόιμπινγκ. Μας είπαν ότι επιτέλους είχε καταπολεμήσει ε, για πολύ καιρό ε, προβλήματα με το Δούναβι είχε ζητήσει να γίνει η αναγκαία μελέτη επιπτώσεων για 33 χρόνια δαπανήθηκαν εκατομμύρια για μελέτες θα ήταν πολύ καλύτερο να έχουν επιλεγεί από πολύ νωρίτερα εναλλακτικέ λύσεις. Καλό παράδειγμα αυτό για το πώς πρέπει να διδακτώ, να, να βγάζουμε συμπεράσματα. Η κυρία Φώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Δύο-τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Συνολικά, κατά τη γνώμη μου, τα κράτη-μέλη έχουν διαχειριστεί σωστά και αρκετά καλά την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και γιατί, γιατί το σύστημα προβλέπει ευελιξία. Όλα τα κρατημέλη έχουν προβλέψει διαφορετικές διαδικασίες, έχουν αναθέσει το καθήκον αυτό σε διαφορετικούς φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και του καθεξής. Στόχος του εγχειρήματο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκολύνει την κατάσταση και γι' αυτό μιλάμε και για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τούτο λεχθέντον όμως μας προσβληματίζει κάπως το περιεχόμενο του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται πολύ ωραίο, σαν μία μονοαπευθυντική θηρίδα. Ωστόσο, είναι πολύ πιο περίπλοκο το περιεχόμενο αυτό και δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όλοι αυτοί οι φορείς να συνεργαστούν και αν πρέπει να περιμένουμε τον ένα να βγάλει ένα πόρισμα για να μπορέσει να συνεχίσει και να πάρει τη σκητάλη ο άλλος δεν θα υπογειωθεί κανένα project ποτέ και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, γιατί να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε 2.700 project τα οποία ε, τα αφορούσε αυτή η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αυτό το οποίο προτείνεται αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ακόμα πιο μικρά έργα να ελέγχονται υπ' αυτή την έννοια. Άρα θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο μισό εκατομμύριο project που θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου για να προχωρήσουν. Είναι γελίο αυτό, εξαιρετικά χρονοβόρο, δαπανε, δαπανηρό και δεν χρειάζεται και τόσο πολύ. Εάν ε, ε, το θέμα είναι μεγάλη αυτή κινητοδρόμη, εάν το θέμα είναι μια μονάδα παραγωγής ε, ε ενέργειας συμφωνούμε. Εάν το θέμα όμως είναι μία απλή παρακαπτήριος γύρω από ένα χωριό, τότε δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσει κατά πόσο υπάρχει περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Οι τοπικές αρχές πρέπει να το κάνουν. Από εκεί και πέρα, σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξουμε αυτή την τάση επέκτασης ε, του πεδίου εφαρμογή, αλλά και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας οι εργολάβοι, οι όλοι οι ανάδοχοι, αυτοί είναι που εργάζονται εκ του σύνεγγυς με τον τοπικό πληθυσμό και με τους τοπικούς φορείς. Ε, σε αυτούς θα πρέπει ε, να δοθεί ε, προσοχή. Συν της άλλης, ως προς τους ειδικούς και εμπειρογνώμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλα μέλη, έχουμε εμπειρογνώμονες που χαίρουν άκρα σεβασμού ε, όταν μιλάτε για διαπιστευμένους, μιλάτε για ένα σύστημα αδειοδότησης ανθρώπων, ε, το οποίο δεν απαιτείται. Αν κάποια θέλουν να προβλέψουν ένα σύστημα διαπίστευσης και αδειοδότησης, να το κάνουν. Αλλά μην αναφέρετε αυτό τον όρο γιατί αποκλείει ε, τα δικά μας συστήματα. Το δικό μας συστήμα, το σύστημα είναι αυστηρό, είναι πολύ καλό, έχουμε τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή που λαμβάνουν τις αποφάσεις. είναι κάτι το οποίο λειτουργεί καλά ήδη και νομίζω ότι δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να μας περιπλέξει τα πράγματα στη δική μας χώρα ε, και να το κάνει δίσκαμπτο και επαχθές. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό. Κατά τα λοιπά θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά του. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αμπατής από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να υπενθυμίσω τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την πρόταση αυτή. Πρώτον, να βελτιωθεί το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, κάτι το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο και, στην, και στον τουρισμό. Δεύτερον, η διαδικασία να ευθυγραμμιστεί, να εναρμονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ε, έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφούνται με τους ίδιους κανόνες, να υπάρχει ένα παιχνίδι επίσης όρης για όλους. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τροπολογίας του εισηγητή εκφράζουμε τη γενικότερη μας ικανοποίηση για τη δουλειά του, ως προς τις τροπολογίες 7 και 10. Κατανοούμε ότι ίσως υπάρχει θέμα εκεί, πράγματι, ε, για τα ε, project στρατηγικού κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να οριστούν πολύ περισσότερα και ως προς την απαγόρευση παράτασης ε, τριών μηνών. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, αλλά ίσως είναι θέμα επικουρικότητας και αναλογικότητας. Η απαγόρευση ενδεχομένως είναι εξαιρετικά ε, αυστηρός όρος στη διατύπωση. Από εκεί και πέρα, ως προς την έλλειψη ευελιξίας και τις υπερβολικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται, κάτι το οποίο έθεσε μόλις τώρα το αξιότιμο μέλος της Επιτροπής σας, ε, η υποχρεωτική ε, ο υποχρεωτικός καθορισμός του πεδίου εφαρμογής ε, εξαρτάται και από τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή καθορίζουμε υποχρεωτικά το πεδίο εφαρμογής στην αρχή και έτσι εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα και από πλευράς αναδόχου ή εργολάβου και από πλευράς δημοσίων φορέων. Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε καλύτερα εάν προκύπτουν θέματα κλιματικής αλλαγής και βιοπικιλότητας και γι' αυτό σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένουμε σε αυτό στον υποχρεωτικό διαφορετικό ε, ε, χαρακτήρα του προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής. Ως προς το 5.3 της πρότασης, οι διαπιστευμένοι ειδικοί υπηρογνώμονες είναι μία από τις δυνατότητες που προσφέρονται στα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η ποιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εθνικές επιτροπές ειδικών. Βεβαίως έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία η δική σας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς ε, θέλουμε ε, να μεριμνήσουμε για την ποιότητα της έκθεσης αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν δεν είναι καλής ποιότητας αυτή η έκθεση, τότε επηρεάζονται οι αποφάσεις που θα ληφθούν από τους αρμοδίους φορείς και θα υπάρξουν και πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες στη συνέχεια. Ίσως ο όρος διαπιστευμένη σημαίνει κόστος για κάποια κράτη-μέλη, έτσι το ερμηνεύουν. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει ευελιξία. Κάθε κράτος μέλος θα μπορέσει να προβλέψει το σύστημα που καλύτερα του ταιριάζει, πάντοτε μεριμνώντας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις εκθέσεις. Ευχαριστούμε κύριε Κουσιέρη, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ήταν πολύ αξιόλογες οι συνεισφορές τους, με βοηθούν, τις σημειώνω και θα τις λάβω υπόψη μου. Ειδικότερα ως προς τις τροπολογίες υπαριθμών 7 και 10, για να μην έχουμε καθυστερήσει στα διάφορα project, ε, είναι αυτό σημαντικό που έχει υποθεί, εγώ είμαι ανοιχτό σε κάθε συζήτηση, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι που μπορείτε να υποβάλλετε για να βελτιώσετε το κείμενο, καταλεκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η Τετάρτη Ιουνίου. Δεν έχετε πολύ χρόνο, δεν έχουμε πολύ χρόνο, άρα παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μου το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω και εγώ στα μέλη ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η τετάρτη. Ιουνίου, Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 18 Ιουνίου. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει ψηφοφορία στις 10 Ιουλίου. Άρα η πρώτη προθεσμία που ατενίζουμε είναι η 4η Ιουνίου για την υποβολή τροπολογιών. Τώρα έχω ένα δίλημα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε προχωρήσει εξαιρετικά γρήγορα και δεν έχει έρθει ο εισηγητής για το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης και δεν έχω και σκιώδεις εισηγητές για τα επόμενα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης. Είχα σκεφτεί να κάνουμε μια ανταλλαγή και να εξετάσουμε πρώτα το κείμενο του κυρίου Δανέλη, αν συμφωνείτε. Και στη συνέχεια ε, την ε, έκθεση Παχνιού. Αλλά αν έχετε αντιρρήσει δεν το κάνουμε. Σας προτείνω λοιπόν να εξετάσουμε την έκθεση του κυρίου Δανέλη πρώτα και την έκθεση Παχνιό μετά. Εάν έχετε αντιρρήσει δεν θα το κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι ίσως ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος να μην είναι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι που καταλαβαίνω. Τι λέτε, συμφωνείτε να εξετάσουμε την έκθεση του κύριου Δανέλη. Πολύ ωραία. Η γαλάζια ανάπτυξη. Σπύρο. Ε, σχετικά λοιπόν με τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφου. δεν έχω πολλά πράγματα να πω. το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν είναι 131 καλύπτουν συνολικά όλο το φάσμα της, ε, των θεμάτων της ε, έκθεσης. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των τροπολογιών, η πολύ μεγάλη, είναι στην κατεύθυνση και στους άξονες ε, και στην λογική της έκθεσης και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσουμε σε συνεργασία στενή με τους σκιώδεις συγητές, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για ολόκληρη τη συνεργασία, ε, να μαζέψουμε τις περισσότερες από αυτές σε 19 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, η προσπάθεια είναι, που έγινε είναι στο να μην κάνουμε πλαδαρό το κείμενο, να μπορέσουμε να το ε, έχουμε όσο γίνεται πιο συγκροτημένο και συνοπτικό. Να πω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών έχει να κάνει με την επισήμανση της μεγάλης προσοχής σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να επιδειχθεί στην προσπάθεια της ανάπτυξης των κλάδων της θαλάσσιας οικονομίας γιατί όλοι αναγνωρίζουμε σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την μεγάλη ευαισθησία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για αναπτυξιακές δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισμός κατεξοχήν το κεφάλαιο που επενδύουμε είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος. Ε, να πω ότι αρκετές τροπολογίες είχαν να κάνουν με τις ε, διατομεακές θαλάσσιες πολιτικές και ιδιαίτερα με τον ολοκληρωμένο θαλάσσιο σχεδιασμό. Η μεγάλη πλειοψηφία των αδέλφων στηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής αυτές. Και επίσης να επισημάνω ότι ε, τα κενά γνώσης αλλά και η ιδιαίτερη ευαισθησία των παρεμβάσεων οι οποίες πρόκειται να εξελιχθούν ε, σε σχέση με την ανάπτυξη του ιδιαίτερου υποτομέα της εξόριξης των ορυκτών και την βιοτεχνολογία ε, είναι οι τομείς τους οποίους ε, επισημαίνεται με πιο έντονο τρόπο αυτή η αναγκαιότητα προστασίας περιβαλλοντικής σε κάθε μας επέμβαση. Να Υπενθυμίσω επίσης ότι πήραμε υπόψη μας ε, δύο γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής ε, Αλληλείας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που και οι δύο γνωμοδοτήσεις ήταν στον, στους άξονες και στη λογική της έκθεσης. Και τέλος ε, να πω ότι επίσης μια, ένα σημαντικός αριθμός τροπολογιών είχαν να κάνουν με την επισήμαση της ιδιαίτερης προσοχής στα ζητήματα της νησιωτικότητας στη διαφοροποίηση δηλαδή των συνθήκων με, τους, με τις οποίες, υπό τις οποίες ε, έχουμε την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας στην νησιωτική περιφέρεια της Ευρώπης από ότι στην υπηρετική. Ε, να ευχαριστήσω θέλω τους ε, συναδέλφους θερμά για την συνεργασία της στενή που είχαμε όπως επίσης και τους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες και με τους οποίους συνεργαστήκαμε στην πορεία αυτή και να ευχαριστήσω τέλο τη Γραμματεία για τη στενή και αποδοτική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δανέλη. Κύριε Κράμερ, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε εξ του ΕΛΚ ή να πάω στην κυρία Μάισνερ. Ξέρω ότι άλλη θα πρέπει να ήταν η ομιλήτρια. Κύριε Κιού. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή είναι πολύ σημαντική έκθεση που απασχολεί, την απασχολεί το πώς θα αξιοποιήσουμε και πώς θα ε, αντιμετωπίσουμε τη θάλασσα. Η μπλε ανάπτυξη έχει να κάνει και με την αυτιλία, με την ενέργεια, με την περιφερειακή, την τουριστική πολιτική, την αυτιλία την ανέφερα ήδη, όλα αυτά να συντονιστούν είναι δυσχερές καθήκον. Ο συνάδελφος Δανέλης, κατά τη γνώμη μου, κατάφερε να τα συνδυάσει όλα αυτά πολύ καλά. Υπάρχουν τροπολογίες, θα τις υποστηρίξουμε. Πολύ σημαντικό για μας είναι να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ξέρετε ποια είναι η οικονομική κατάσταση σε πολλές από τις χώρες μέλη, ιδιαίτερα δυσχερείς, ε, Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ανάπτυξη λοιπόν, να προωθηθεί ανάπτυξη και φυσικά και ο θαλάσσιος τομέας είναι πολύ σημαντικός και υποστηρίζουμε την προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Σπύρο Δανέλη. Θαυμάσια εργασία, πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ των σκιωδών και του εισηγητή. Όπως είπε ο κύριος Κούν, η μπλε ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική με από το ίδιο ομοσπονδιακό κράτος με την κυρία Μέρκελ είπε ότι οπωσδήποτε η κυρία Μέρκελ ε, η θαλάσσια πολιτική θα παίξει μεγάλο ρόλο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα βεβαίως η ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική και η γαλάζια ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και για την στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρέπει να συνδυαστούν λοιπόν αυτά τα δύο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην ε, Μάλτα για την Ευρωπαϊκή ημερίδα θαλασσών ως ε, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφέρθηκα στην έκθεσή μας, αναφέρθηκα στις προσπάθειες που κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο δυναμικό σε αυτό το τομέα και κάτι άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα και με ε, φοιτητές στο Bremerhaven και ε, με ρώτησαν πόσο μας απασχολεί η βιωσιμότητα στη θαλάσσια πολιτική και τους είπα ότι είναι βασικός τομέας αυτός, βασική προημόθεση γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θάλασσα εάν πραγματικά ε, φροντίσουμε να προστατευτεί το περιβάλλον. Αυτός είναι λοιπόν ο πυρήνας. Δεν έχω πολλά να πω για τις τροπολογίες. Χθες καθίσαμε μαζί, συζητήσαμε τις συμβαστικές τροπολογίες και ε, σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε ε, από πλευρά μου, εκτό από δύο συμβαστικέ τροπολογίε, θα υποστηρίξουμε όλε τι άλλε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κύριε Φώστερ έχετε εντολή να μιλήσετε εξ ονόματος του κύριου Ζήλερ. Σας δίνω το δικαίωμα αν θέλετε. Όχι, ο Πίτερ Βαντάν ήταν νομίζω ο σκιώδης ηγητής. Είχαμε διάφορες παρατηρήσεις να κάνουμε, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες βεβαίως, γιατί ο Πίτερ είναι ο επίσημος σκιώδης εισηγητής. Θεωρούμε όμως ότι όλα αυτά ε, προδιαγράφουν με υπερβολικό βαθμό τις ε, δυνατότητές μας. Η νομοθετική προσέγγιση μας, μας προβληματίζει και όχι τόσο η εταιρική, αν θέλετε. προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας, αυτά είναι καλά. Ε, όχι όμως τόσο στο νομοθετικό επίπεδο. Θέλουμε σε νομοθετικό επίπεδο να υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο, καλό, μέσα στο οποίο, μέσα στο οποίο τα κράτη-μέλη να μπορούν να δουλέψουν. Δεν θέλουμε το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια όλους τους κανόνες. Βεβαίως θα εξετάσουμε τις τροπολογίες Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πράγματι έχει κάνει πολλή δουλειά. Δεν είναι ότι δεν θέλετε την βιώσιμη ε, ανάπτυξη. Και εγώ από νησί ε, είναι η καταγωγή μου. Ξέρω ότι και εσείς το ίδιο επιθυμείτε. Το θέμα είναι ε, ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είμαι πεπισμένη ότι είναι αυτή η σωστή προσέγγιση του προσδιορισμού των πάντων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, έχετε δίκιο, ο Πίτερ Βαντάντε είναι ο σκιώδης συζητητής εξ ονόματος του ECR. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό γιατί είναι πολύ νωρίς, το είχαμε προγραμματίσει αυτό το σημείο για αργότερα. Κύριε Δαντέλη, έχετε κάτι να προσθέσετε. Μονάχα ε, δύο κουβέντες, μία επισήμανση κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στις, στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι ε, η απώλεια της ανταγωνιστικότητας σε σχεδόν όλους τους τομείς και η μεταφορά του κέντρου οικονομικής ισχύω ε, ανατολικότερα και νοτιότερα της Ευρώπης. Νομίζω ότι όπως τώρα και 7.000 χρόνια ή και περισσότερο οργανωμένα οι παππούδες μας, οι προπαπούδες μας στην Ευρώπη ε, αναζητούσαν την ε, όχι μονάχα τη διαβίωση, την επιβίωση, αλλά και την ανάπτυξη ε, στρεφόμενη στη θάλασσα, έτσι και σήμερα είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση, αναζητώντας τη χαμένη ανταγωνιστικότητα η Ευρώπη να στραφεί στη θαλάσσια οικονομία. Γνωρίζει πολύ καλά τους δρόμους, καλύτερα από οποιονδήποτε, και όλοι οι τομείς οι οποίοι αναφέρονται στην ε, ανακοίνωση Επιτροπής για την γαλάζια ανάπτυξη νομίζω ότι είναι ε, τομεί του οποίους η Ευρώπη διαθέτει ε, πλεονεκτήματα σημαντικά και βεβαίως ε, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και η απάντηση σε ένα μεγάλο κομμάτι της κρίσης και στην οικονομία αλλά και της μεγάλης κοινωνικής κρίσης για τη δημιουργία πολύ μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας. Είναι οραματικό και φιλόδοξο το σχέδιο αλλά ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστικό. Ευχαριστώ ξανά τους συναδέλφους σκιώδες ηγητές αλλά και τους συναδέλφους που βοήθησαν στην διαμόρφωση της τελικής έκθεσης όπως επίσης και τη γραμματεία και τους συνεργάτες του γραφείου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δανέλη. Κύριε Τέιλορ. Μήπως να αλλάξουμε λίγο τα σημεία της ημερήσιας ε, διάταξης. Ξέρω ότι μόλις ήρθατε. Θέλετε να πείτε κάτι για την έκθεση Δανέλη. Έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Τέιλορ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν συντομία να πω Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μπόρεσε να πάρει υπόψη του τόσες, τόσες πολλές ε, καλές προτάσεις στις συμβαστικές ε, προτάσεις που υπέβαλε ο ίδιος. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία σε σχέση με τις ε, οικονομικές δραστηριότητες και άλλες θαλάσσιες αυτό δυστυχώς δεν το ε, πετυχαίνει η πρόταση της Κομισιόν στα πλαίσια της γαλάζιας ανάπτυξης. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή η κατάλληλη ισορροπία σε σχέση με την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτή καθεαυτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Τέλος πάντων, ε, για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, εγώ πιστεύω ότι η κατευθυντήρια γραμμή η βασική πρέπει να είναι βιωσιμότητα βιωσιμότητα της γαλάζιας ανάπτυξης και μια κατάλληλη εφαρμογή, αναγνώριση και εφαρμογή της αρχής της σύνεσης όπως εμφανίζεται και στην συνθήκη. Η οικονομικές δραστηριότητες δεν πρέπει να ε, ε, αποκτούν προτεραιότητα σε σχέση με, την, ε, με το θαλάσσιο περιβάλλον και την υγεία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει συνεργασία διότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αναγκαστικά και ομοιόμορφοι και ενιαίοι κανόνες κάτω από οποιαδήποτε συνεργασία συνθήκες. Ε, υπάρχουν ναυάγια τα οποία λαμβάνουν και, ε, ε, και η, καταστροφή των πλοίων ε, γίνεται κάτω από περίεργες και, και διαφορετικές συνθήκες. Επομένως όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται με πολύ σοβαρό τρόπο και Ούτως ή άλλως εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αναπτυχθεί ο βιώσιμος τουρισμός ταυτόχρονα. Ε, η συμβαστική πρόταση 5 και 16 δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι λάβατε υπόψη σας και δεχτήκατε αυτές τις ε, αλλαγές που κάναμε στην μερίσια διάταξη. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία είναι αύριο και να καλωσορίσω επ' ευκαιρία τους 16 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Κάσελ που έχουμε μαζί μας, είναι στην, στο βάθος της αίθουσας. Η κυρία Βέιλερ τους προσκάλεσε από τους σοσιαλιστές και σας καλωσορίζουμε και ελπίζω να βρήκατε κάπως ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις. Είμαστε, σήμερα το πρωί μας απασχολεί το θαλάσσιο περιβάλλον, ε, πλέουμε στα κύματα του ωκεανού. Σας καλωσορίζω πάντως. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την έκθεση του κυρίου Παγνιό για τα φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από τις 26 Απριλίου που ήταν η τελευταία προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών ήρθα σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές για να βρούμε κάποιες συμβιβαστικές ε, προτάσεις που θα διευκολύνουν την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα αύριο στην Επιτροπή μας. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές ε, για την κατανόηση που έδειξαν όταν προσπαθούσαμε να συντάξουμε αυτές τις συμβιβαστικές προτάσεις οι συμβιβαστικέ προτάσεις αφορούν τα άρθρα 11, 13, 19 και το παράρτημα 5. Η ολοκληρωμένη τροπολογία 2 αφορά το άρθρο 11.3 και καλύπτει τις τροπολογίες 19, 77, 82 και την αιτιολογική έκθεση 7. Η τροπολογία αυτή μας επιτρέπει να επιτρέψουμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2003 την ε, συντήρηση και την διατήρηση των ψυκτικών μηχανισμάτων, μηχανημάτων που, συμπερι, που περιέχουν φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου. Και ε, επιτρέπουμε δηλαδή στους κατασκευαστές ψυγείων που έχουν πρόσφατα επενδύσει ε, στον εξοπλισμό, τον να διατηρήσουν την, τα μηχανήματα των εξοπλισμό τους και να προσαρμοστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και εδώ συμμετέχουν αρκετές πολιτικές ομάδες. Η ολοκληρωμένη ε, τροπολογία 2 αφορά το άρθρο 13 παράγραφος 4.1 και καλύπτει τις τροπολογίες 93 και 94. Η τροπολογία αυτή μας επιτρέπει να ε, επιμένουμε ε, στην, την, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα των φθοριωμένων αερίων αλλά θα πρέπει και η Κομισιόν να φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει στην αγορά διαθέσιμη μια εναλλακτική λύση ε, που θα είναι από τεχνικής και οικονομικής πλευράς βιώσιμη. Ε, η πρόταση αυτή γίνεται δεκτή από την ΚΟΕ, από τους πράσινους, από τους σοσιαλιστές κτλ. Η τροπολογία 3 ε, αφορά την ε, παράγραφο 10, το άρθρο 19, 3 και καλύπτει τις τροπολογίες 23 και 115. Η τροπολογία αυτή αφορά, προ, αφορά και μια προστιθέμενη αξία της ε, οδηγίας ε, που, μας, ε, που θα κυκλοφορήσει στην, στην ευρωπαϊκή αγορά αν θέλετε. Η οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2022 και το 2024. Η έκθεση αυτή επίσης θα συμπεριλαμβάνει και κάποιες ε, απαιτήσεις για, ε, για υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την χρήση των φθοριούχων αερίων το 2024 και μετά το 2030 τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 4 αφορά την, ε, το άρθρο 5, ε, αφορά τις τροπολογίες 29, 30 και 130, 135. Ε, και εδώ ορίζεται η μέγιστη ποσότητα των φθοριωμένων αερίων που η παραγωγή και η εισαγωγή μπορούν να κυκλοφορήσουν στην κοινοτική αγορά κάθε χρόνο. Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων, οι θέσεις των μεν ήταν ε, ριζικά αντίθετες από τις θέσεις των δε πάρα πολλές φορές. Όμως καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική πρόταση που ορίζει ε, στόχους φιλόδοξους αφήνοντας όμως παράλληλα και τον απαραίτητη χρονική περίοδο προσαρμογής για την βιομηχανία. Η τροπολογία αυτή είναι συμβιβαστική και την ε, ε, υποστηρίζει το ΕΛΚ οι σοσιαλιστές μεταξύ άλλων. Επίσης να σας υπενθυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι θα ψηφίσουμε το κείμενο αυτό αύριο, γύρω στις 9 και 10. Ε, πιστεύω και εγώ ότι θα το ψηφίσουμε τότε. Αλλά η δυνατότητά μου σήμερα να τηρώ το πρόγραμμα έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Αλλά η ψηφοφορία θα γίνει αύριο για το ΕΛΚ. Κύριος Μπάνκι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παγνιό για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μαζί του. Το ανέφερε και αυτός στην εισαγωγή του. Ήταν πολύ αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Υπήρξαν σημεία που είχε προτείνει το ΕΛΚ και που με χαρά διαπίστωσα ότι λήφθηκαν υπόψη. Υποστηρίζουμε λοιπόν την απαγόρευση αυτών των φθοριούχων αερίων όταν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι επικίνδυνα αυτά τα νέα προϊόντα και να μην σημαίνει η εισαγωγή τους και τεράστια αύξηση του κόστους. Πρέπει να τονίσω ότι από πλευράς της Τραν το θέμα αυτό τα αέρια που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ψυκτικές εγκαταστάσεις, ε, σε φορτηγά ψυγεία κτλ. Θέλουμε λοιπόν όλος αυτός ο τομέας, αυτό το τομέα ακριβώς θέλουμε να τον βγάλουμε από την ε, ε, πρόταση αυτή, όπως και για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος γιατί για τους τομείς αυτούς ε, δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσεις που θα τηρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Οι συμβασμοί λοιπόν, που αναφέρθηκαν ε, μπορούν να υποστηριχθούν σε τρεις περιπτώσεις από το ΕΛΚ, ε, σε τρεις περιπτώσεις έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία που βελτιώνουν το κείμενο. Με τον δεύτερο συμβασμό έχουμε προβλήματα γιατί Το ΕΛΚ θα ήθελε να είναι πιο αυστηρές ε, οι προδιαγραφές, αλλά να υπάρξουν και απλούστερες ρυθμίσεις. Ορισμένα αέρια δεν μπορούν να ε, εξαιρεθούν, αλλά σε άλλες περιπτώσεις ε, θα έπρεπε να δούμε πώς συνδυάζονται οι βιομηχανικές αλλά και οι μορφές ασφαλείας. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Παγνιό για την εργασία, για την καλή συνεργασία. Είναι σημαντικό να αντικατασταθούν αυτά τα αυθοριούχα αέρια γιατί συμβάλλουν περισσότερο από το διοξίδιο του άνθρακα στην ε, θέρμανση του πλανήτη εδώ θέλουμε να καταπολεμήσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, άρα και αυτά το θέμα είναι τι εναλλακτικέ λύσεις έχουμε. Δεν έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι δύσκολο να τα υποκαταστήσουμε, γιατί ορισμένες εναλλακτικέ λύσεις είναι ιδιαίτερα έφλεκτες. Ε, ορισμένα πολύ έφλεκτα, ορισμένα μετρίως έφλεκτα, άρα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Γενικά, όπως είπε και ο εισηγητής, υπάρχει ευρεία συνένεση. Θα υποστηρίξουμε όλοι τις συμβαστικές τροπολογίες. Πρέπει όμως να σκεφτούμε εάν ε, έχουμε ήδη ε, έχουμε ήδη παντού εναλλακτικέ λύσει. Για παράδειγμα, για τον κλιματισμό των ε, τρένων, όπω είπε και ο συγκητή του ΕΛΚ, δεν έχουμε πάντα εναλλακτικέ λύσει. Άρα πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσει. Θα ζητήσει η ομάδα του. Επίση για το διάστημα και για τον τομέα τη υγεία. Θα τα υποστηρίξουμε και εμεί αυτά. Αλλά κατά τα υπόλοιπα είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτό το τομέα. Ο, για όλα όσα αφορούν βεβαίω ε, τις μεταφορές που μας ενδιαφέρουν. Ο κύριος Τέιλορ για του πράσινου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παγνιό για τη δουλειά του. Νομίζω ότι επέδειξε πνεύμα πραγματικής ε, συνεργασίας είχε τη βούληση να προχωρήσουμε πράγματι ε, σε αυτή την έκθεση, να αναλάβουμε φιλόδοξη δράση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Στον οδικό χάρτη ε, για να προχωρήσουμε σε μια ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα το 2020. Υπήρχε αυτή η ευκαιρία, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ε, την έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Ο τομέας των μεταφορών έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι πολύ φιλόδοξη ως προς την ε, μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και τον, ως προς τη μείωση της χρήσης των φθοριούχων αερίων. Δεν χρειαζόμαστε περιττέρω έρευνα. Έχουμε τη γνώση. Πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να μειωθούν αυτά τα επίπεδα και υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις στους περισσότερους τομείς. Η φιλόδοξη δράση είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν τις τεχνολογίες αντικατάστασης, υποκατάστασης αυτών των ε, προϊόντων με άλλα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Δυστυχώς, οι πολυεθνικές είναι αυτές που προωθούν τα CFC, τα οποία παράγονται και στην Κίνα κιόλας. Ε, δουλέψαμε πολύ, προσπαθήσαμε πολύ να βρούμε συμβαστική λύση για την τροπολογία υπαριθμών 4. Η έλλειψη φιλοδοξίας δεν το κατέστησε αυτό εφικτό. Επομένως δεν θα υποστηρίξουμε την τροπολογία υπαριθμών 4. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φώστερ, είστε πράγματι αρμόδια να μιλήσετε εξ ονόματος του κυρίου Ζήλερ, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι έχει χαθεί κάπου. Ε, θα είχε τα δικά του σχόλια να κάνει, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τους κοιόδες εισηγητές για την δουλειά τους. Πράγματι έχουν κάνει σκληρή δουλειά. Είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεση αυτή. Δεν νομίζω ότι είμαστε χημική εδώ και γνωρίζουμε τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε με τι, όλα αυτά μου θυμίζουν λίγο το τι γινόταν με τον κανονισμό REACH, το οποίο μας είχε τρελάνει όλους και είναι κάτι που εκτιλισόταν για χρόνια ολόκληρα. Τώρα θέλουμε τη σταδιακή εξάλληψη των φθοριούχων αερίων. Εν πάση περιπτώσει, για κάποια από τα άρθρα που έχουν τροποποιηθεί με τις τροπολογίες, ε, εμείς θα τα στηρίξουμε. Θεωρούμε ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το άρθρο 8 για την κατάρτιση, για την πιστοποίηση, ε, το 11 ε, υπάρχει εκεί συνένεση για το έβρος του κατοφλίου. Το 13 πρέπει να δουλευτεί περισσότερο. Είναι δύσκολη η σταδιακή εξάλληψη, αυτό είναι σίγουρο και το άρθρο 18 αναφέρεται στη συλλογή των δεδομένων για τις εκπομπές και τα συστήματα υποβολής αναφορών. Όλα αυτά είναι συζητήσιμα και πολύ δύσκολα, αλλά εν γενικώς θα μπορούσαμε ίσως να τα υποστηρίξουμε. Αυτό το οποίο μας δημιουργεί τεράστια, ε, τεράστιο πρόβλημα είναι η ενδυνάμει απαγόρευση για νέα προϊόντα και η νέα εναλλακτική ε, για το μητρό, ε, για τις ποσοστώσεις και την προκαταβολική απαγόρευση. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουμε να υποστηρίξουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες 1 και, 1 και 2, αλλά όχι την 3 και 4 και όχι όλες αυτές οι ημερομηνίες και τα ποσοστά. Τα ποσοστά με προβληματίζουν, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά η Επιτροπή έχει καταλήξει σε ποσοστά μεταξύ συγκεκριμένων ημερομηνιών, τα οποία είναι τόσο συγκεκριμένα και αυτά που δεν μπορώ να την πιστέψω πια. Δεν λέω να μην θέτετε στόχους, αλλά να προβλέπετε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο 63% ή στο 31% και όχι στο 32% ή στο 30% αυτό είναι ένα τέχνασμα, είναι κάπως περίεργο. Καλή την πίστη πρέπει να λειτουργούμε. Είναι καλύτερα αυτά τα νούμερα από άλλα που δεν έχουμε ή που δεν γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να δουλέψουμε ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και θα πρέπει να το δούμε το θέμα και με την Επιτροπή ΕΜΒΗ. Σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, ε, το, η σταδιακή εξάλληψή μας δημιουργεί προβλήματα, η αντικατάστασή μας δημιουργεί προβλήματα. Όλα αυτά φαίνονται ομαλά εκ πρώτης όψεως, αλλά δεν είναι. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει το όλο αυτό το θέμα και χωρίς τη δική μας συνεισφορά. Κατά τα λοιπά ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Βίλς. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει σταδιακή μείωση, face down, και δεν είναι οι ποσοστώσεις αρκετά αυστηρές. Τα αέρια αυτά είναι βλαβερά, χρειάζονται απαγορεύσεις, όχι μείωση. Θέλω και έχω εισαγάγει τροπολογίες για την απαγόρευση. Πρέπει να αντικατασταθούν τα αέρια αυτά σε ορισμένους τομείς είναι δυνατόν το 2015, σε άλλους το 2020 και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη προθεσμία. Είναι απόλυτα εφικτά όλα αυτά. Τώρα επιδιώκεται περαιτέρω αποδυνάμωση των διατάξεων. Ξέρετε ότι οι παραγωγοί αλλάζουν την παραγωγή τους μόνο εάν υποχρεωθούν πρέπει να εισαχθούν απαγορεύσεις για να υπάρξει σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι πρέπει να αναλάβουν τις αναγκαίες επενδύσεις και αλλαγές στον τρόπο παραγωγής τους. Όταν υπάρξει η απαγόρευση, τότε μόνο οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την προσφορά τους στη ζήτηση. Όλοι αυτοί που είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς θα πρέπει να τα καταλαβαίνουν αυτά. Έτσι συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επιτρέπουμε και στις επιχειρήσεις μία ασφάλεια στα επιχειρηματικά του σχέδια. Οι απαγορεύσεις έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν δεν έχουν ατελείωτα παραθυράκια μέσω εξαιρέσεων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα ε, μάλλον να μην δώσουμε στα κράτη-μέλη τη, τη, δυνατότητα να εισάγουν εκείνα παραθυράκια Πρέπει να βρούμε κοινή θέση, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κανονισμός έχει έννοια μόνο εάν κλείσουμε όλα τα παραθυράκια και σκεφτούμε λογικά και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κυρία Βίλς για την Επιτροπή. Ο κύριος Ράιν, νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει στις θαλάσσιες οδούς. Ο κύριος Ράιν από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση και για, την ε, συζητή και για τις συζητήσεις. Δεν μπορώ βέβαια να σχολιάσω το περιεχόμενο των συμβαστικών, τροπολογιών γιατί δεν το έχουμε, το έχουμε δει ακόμα. Αλλά τέλος πάντων, επί της αρχής σχετικά με τα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί εκτενώς παραδείγματο χάρη για τις ε, υπηρεσίες και την απαγόρευση και για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής ε, των σχετικών διατάξεων. Θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να ε, υπενθυμίσουμε ότι το ε, η θετική επίπτωση στο περιβάλλον και εξαρτάται και από την ημερομηνία που θα είναι ε, αποτελεσματική η απαγόρευση. Τώρα όσον αφορά αυτό το phased out, πρέπει να εξηγήσω γιατί καταλήξαμε σε τόσο συγκεκριμένα ποσά και ποσοστά και πώς ε, υπευλήθη η πρόταση αυτή έγινε με βάση μια συγκεκριμένη μελέτη που μελέτησε, που εξέτασε τις ε, απαιτήσει και, ε, και που έλαβε υπόψη την, ε, την οικονομική και την εμπορική και την περιβαλλοντική πτυχή της παροχής ασφαλούς ενέργειας. Όταν δημιουργείς ένα χρονοδιάγραμμα με βάση κάποιο μοντέλο, θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και να ε, παραμένεις πιστός, αν θέλεις, στο αποτέλεσμα. Λάβαμε υπόψη μας το 60, διότι το 63 θεωρήσαμε ότι δεν θα ήταν τόσο αξιόπιστο Επομένως, μπορείτε να δείτε εδώ κάποια περίεργα στοιχεία, περίεργα ποσοστά, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι έχουμε υιοθετήσει μια ιδιαίτερα συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν και την τεχνολογία και αυτό το οποίο μας δημιουργεί είναι να ε, διατηρήσουμε την ασφάλεια, τα περιθώρια ασφάλειας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εναλλακτική τεχνολογία προχωρά πάρα πολύ γρήγορα αν λάβουμε υπόψη μας ε, τι στοιχεία είχαμε το 2008 όταν ξεκινήσαμε την μελέτη, θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα και διαθεσιμότητα σήμερα. Επομένως, δημιουργήσαμε κάποια περιθώρια ασφάλειας στην έκθεσή μας και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας όταν συζητάμε ε, το όλο πρόγραμμα περιοδικής ε, μείωσης. Ε, κύριε Παγνιό, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των σκιωδών εισηγητών και τις ομάδες τους για τη δουλειά που έχουν κάνει Πιστεύω ότι όπως ε, το θυμήσατε και όλοι σας ε, καταφέραμε να βρούμε αυτή την ευαίσθητη ισορροπία. Από τη μια πλευρά υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε για να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές ε, συνέπειες και επιπτώσεις των φθοριωμένων αερίων. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να επιτρέψουμε στην βιομηχανία, στον κλάδο αυτό, να λειτουργήσει όπως πρέπει σε μία, μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας ε, η οποία περνάει κρίση. Σε αυτές τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, ε, κυρίες τις συμβαστικές τροπολογίες 3 και 4, σε σχέση με αυτά που είπατε κυρία, κυρία Φώστερ, είχε επιτευχθεί μια συμφωνία με τον κύριο Ζήλερ, αλλά ξέρω με, την, με, το, με την ομάδα ECR, αλλά ξέρω ότι και στο εσωτερικό της ομάδας σας δεν ε, είναι όλα τα μέλη στο ίδιο μήκο κύματο ε, σε σχέση με αυτές τις δύο συμβαστικές ε, τροπολογίες. Και αναφέρομαι στους Βρετανούς συντηρητικούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο το πρωί όταν ψηφίσουμε. Τώρα, μπορώ, μπορούμε να, επιτρέψουμε, να επιστρέψουμε συγγνώμη, στη γαλάζια ανάπτυξη και η κυρία Βλαστό ήρθε δεν έφταιγε εκείνη επειδή αλλάξαμε εμείς την σειρά των ε, σημείων της ημερήσιας διάταξης και είχα ε, ε, υποσχεθεί στην κυρία Βλαστό ότι θα μπορείς να κάνει ε, μια τέτοια παρέμβαση εδώ σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καθυστέρησα λόγω τρένου και ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να ε, ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας ε, για τη δουλειά που έκανε και γιατί μας άκουσε και επίσης ε, και μας επέτρεψε να βρούμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις για κάποια σημεία και αυτό μου, δίνει, μου δημιουργεί μια εμπιστοσύνη όσον αφορά την συνένεση που θα μπορέσουμε να πετύχουμε αύριο στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Όμως θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτές στην έκθεση.

πρέπει να ε, επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό υπάρχει και η αρχή της σύνεσης και η απέτηση να ε, διασφαλιστεί η θαλάσσια ασφάλεια. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε ένα υγιές οικοσύστημα έτσι ώστε να μπορεί να είναι και παραγωγικό. Εξού και χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη για την γαλάζια ανάπτυξη έτσι ώστε να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν δραστηριότητες συντήρησης και ανάκαμψης του ε, θαλάσσιου και παραθαλάσσιου αν θέλετε ε, περιβάλλοντος και κληρονομιάς μας. Ήθελα επίσης να, να πω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποτελεί μια, ένα φύλλο πορείας για, για το κοινοβούλιο μας έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η γαλάζια ανάπτυξη η οποία μας απασχολεί εδώ και καιρό. Πρέπει όμως να τονίσω ότι το ΕΛΚΑ δεν πρόκειται να υποστηρίξει τις τροπολογίες που υπέβαλε ο κύριος Μπιζότο ε, γιατί θεωρούμε ότι την οικονομική κρίση την αντιμετωπίζει με κάποιο ακραίο τρόπο και στηρίζεται με όσα γεγονότα. Η κρίση επηρεάζει όλους τους τομείς, ακόμα και τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας. Όμως θα πρέπει η έκθεση αυτή να αποτελέσει ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο θα μας επιτρέψει να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο για να πετύχουμε την ανάπτυξη. Και έχουμε συμφωνήσει επίσης και με τον εισηγητή να μην υποστηρίξουμε κάποιες τροπολογίες, είτε γιατί θεωρούμε ότι είναι περιτές, είτε γιατί πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς. Αντίθετα, όμως το ΕΛΚΑ υποστηρίζει τις τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των νησιωτικών περιοχών και των απομακρυσμένων περιφερειών ε, και ε, που ε, υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, της αλίας, τέλος πάντων τομέων που επιτρέπουν την γαλάζια ανάπτυξη. Αυτά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Βλαστό. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το... το τέταρτο, η τέταρτη δέσμαση μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και έως. Περιμένω τους πρώτους εισηγητές, κυρία Μπιλμπάου και κύρι, κύριο Ζήλερ, να κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 10.45. Ε, 11 παρατέταρτο λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τέταρτη δέσμη για τους σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε, αγαπητοί συναδελφοί, για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αυτή τη ε, δέσμη για το σιδηροδρομικό χώρο, η οποία δεν εγκύρει και πολλές αντιρρήσεις. Να σας πω πώς θα οργανώσουμε τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με τη διαλειτουργικότητα, μετά την ασφάλεια και μετά τον ευρωπαϊκό ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο. Μετά τη διαλειτουργικότητα θα ακούσουμε τον εισηγητή, τους κοιόδης εισηγητές και μετά τα μέλη. Για την ασφάλεια το ίδιο και για το ERA το ίδιο επίσης. Δηλαδή αναθεματική ενότητα θα συζητούμε για να αποφύγουμε ένα πηδάμα από το ένα θέμα στο άλλο. Και το ίδιο σύστημα θα ακολουθήσουμε και σήμερα το απόγευμα με τις άλλες τρεις υποθέσεις που πρέπει να εξετάσουμε μια μισή ώρα περίπου, 30 λεπτά για κάθε θέμα, να το έχετε υπόψη σας. Ξεκινούμε με τη διαλειτουργικότητα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει γίνει διάγνωση της κατάστασης με βάση τα έγγραφα υποστήριξης που μας έχουν υποβάλει διάφοροι φορείς. Σε 18 συνεδριάσεις που έχουμε οργανώσει μέχρι σήμερα το έχουμε κάνει αυτό και θα έχουμε και άλλες συνεδριάσεις και συσκέψεις τις επόμενες ημέρες. Καταρχάς να πω ότι οι μεταφορές στην Ευρώπη σίγουρα μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο καθαρές, πιο χρήσιμες και πιο φθηνές για τους χρήστες. Ε, προβάλλοντας περισσότερες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες εάν ο σιδηρόδρομος ανοιχτεί στον ελεύθερο ανταγωνισμό και υπάρξουν περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης και μεγαλύτερη και περισσότερη προσφορά. Για όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε το πρόβλημα έλλειψης ε, διαφάνειας. Έχουμε 11.000 ε, διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη-μέλη με την ύπαρξη φυσικών ιστορικών μονοπωλίων και τεχνικών εμποδίων για, την, για το άνοιγμα της αγοράς και θα μπορούσαμε να τα συσχετίσουμε όλα αυτά με την έλλειψη διαφάνειας και ξεκάθαρης κατάστασης. Όλα αυτά εμποδίζουν νέους φορείς εκμετάλλευσης να μπουν στην αγορά, ε, είναι πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, ουσιαστικά δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός και δεν μπορούν να γίνουν σωστές επενδύσεις. Αποθαρρύνονται και έτσι καταραίουν οι κατασκευαστές, οι επενδυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις 11 ολόκληρα χρόνια διαρκούν οι διοικητικές διαδικασίες, κάτι το οποίο είναι τεράστιο πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα και άρα δεν μπορεί και ο κλάδος να επενδύσει. Θα επενέδυε πολύ πιο αποφασιστικά αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά. Τι να κάνουμε. Πρώτον, με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Shift to Rail, αυτή την πρωτοβουλία, τα πορίσματά του να τα ενσωματώσουμε στη δουλειά μας να επιβάλλουμε τη διαφάνεια για τη διαλειτουργικότητα και την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων, να εξαλείψουμε αργά ή μάλλον, σταθερά αλλά γρήγορα τους εθνικούς κανόνες που, που δημιουργούν προσκόμματα, να καθορίσουμε διαδικαστικά πρωτόκολλα για να υπάρξει σαφήνεια, ευκρίνεια, διαφάνεια, ενοποιημένοι κανόνες να υπάρξουν, αποφεύγοντας την ύπαρξη νέων κανόνων και τέλος, να καθορίσουμε σαφέστατα τον ρόλο του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και των ε, κρατικών φορέων. Ποια αποτελέσματα θα πετύχουμε έτσι. Θεωρούμε ότι θα πετύχουμε την πλήρη διαλειτουργικότητα, θα βελτιώσουμε τις συνθήκες για να υπάρξει επένδυση, περισσότερες επενδύσεις στον τομέα, θα ανοιχτεί η αγορά και θα βελτιωθεί η υπηρεσία που προσφέρεται στους χρήστες από πλευράς τιμής, ποιότητας και ασφάλειας. Πώς θα τα πετύχουμε. Έχουμε ιδέες και μάλιστα πολλές. Θα προτιμούσα να ακούσω τους άλλους εισηγητές, να δω εάν συμφωνούμε όλοι με την αποτίμηση της κατάστασης και τα μέτρα που δέον είναι να ληφθούν. Συμμεριζόμαστε λοιπόν τη διάγνωση αυτή, ε, συμφωνούμε με το πρόβλημα συμφωνούμε με τα μέτρα που θα πρέπει να, λυθούν για να, να απαρθούν συγγνώμη, για να λυθεί το πρόβλημα, να δούμε αν όντως ισχύουν όλα αυτά, αν όντως υπάρχει πεδίο συμφωνίας, να δούμε σε ποιο χρόνο και σε ποιο διάστημα θα πρέπει να αναλυφθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και να εφαρμοστούν τα διάφορα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μοιραστούμε τις απόψεις μας για το κατά πόσο συμφωνούμε για το, την εικόνα της κατάστασης και κατά πόσο συμφωνούμε για το τι μέλη και τι δέον γενέστε. Εδώ, σήμερα, στο άρθρο 1, από εκεί και πέρα, είναι πολύ σημαντικό να μην επεκταθεί το πεδίο των εξαιρέσεων. Το 54 πρέπει να μείνει ως έχει, αναφορικά με τους πίνακες συσχετισμών και θα είναι ανάγκη πράγματι να προχωρήσουμε, να γίνει κάτι, ώστε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τη δέσμη των αποφάσεων για το σιδηροδρομικό χώρο, για όλες αυτές τις δέσμες μέτρων και αποφάσεων, γιατί δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Κάθε μία από τις δέσμες μέτρων που έχουν παρουσιαστεί ε, βασίζεται ε, σε δουλειά που έχει γίνει εκ των προτέρων και δεν θα πρέπει αυτή να τη θέτουμε στο περιθώριο. Οικοδομούμε ε, μια Ευρώπη πολύ σημαντική, θα πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση να καταστήσουμε την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική, να δημιουργήσουμε ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης με περισσότερη και μεγαλύτερη καινοτομία. Να πετύχουμε πραγματική διαλειτουργικότητα και έναν ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Σήμερα με τη συζήτηση που θα έχουμε και με τις εκθέσεις που θα εξετήσουμε πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ή αν θέλουμε να διατηρηθεί το status quo, δηλαδή τα μονοπόλια, η κλειστή αγορά και να προβάλλονται τα επιχειρήματα της κρίσης. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς η κρίση λειτουργεί ως επιχείρημα πιστικό για να προχωρήσουμε, για να επιλύσουμε τα προβλήματα που είναι γνωστά σε, όλα, σε όλους έχουν τεθεί επιτάπητος εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει να πάρουμε την πολιτική απόφαση για να φθηνίνει η υπηρεσία, να αυξηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητά της, να χαίρει περισσότερης και μεγαλύτερης διαφάνειας. Κατά τα λοιπά, Τις επόμενες μέρες θα δουλέψουμε πάνω στις λεπτομέρειες, αυτό είναι βέβαιο. Αυτή τη στιγμή, για αυτή τη μια μισή ώρα, θα ήθελα να ακούσω τα άλλα μέλη της Επιτροπής και θα ήθελα σήμερα να αποφασίσουμε αν όντως συμφωνούμε όλοι για την εκτίμηση της κατάστασης, για το πώς έχει η κατάσταση και ποια μέτρα πρέπει να ε, ληφθούν. Αυτά προς το παρόν, ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ την κυρία Μπιλμπάου. Έξι λεπτά για τους εισηγητές, τέσσερα λεπτά για τους σκιώδεις και δύο λεπτά για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Γκρόσφορ είναι ο πρώτος σκιώδης εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, ζητάω συγγνώμη από πλευρά του συναδέλφου Ντεγκράνης το θέμα της απασχόλησης συνολικά για το ΕΛΚ. Ε, ε, μας απασχολεί, όπως είπα, και αν μιλήσουμε χωριστά για την τεχνολογία, παρόλα αυτά αποτελεί τμήμα ενός συνολικού πακέτου και συνδέεται με την συνολική συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και την υποδομή που χρειάζονται. Είμαστε πεπισμένοι εδώ και καιρό, εμείς ως Κοινοβούλιο, ότι οι διαφορετικές τεχνολογίες είναι σημαντική τροχοπέδη στη δημιουργία ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς. Και με αυτά που έχουμε συζητήσει εδώ σε Επιτροπή με τους συναδέλφους. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι ένα τρένο που πάει από το Παρίσι στην ε, Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ηλεκτρική τάση τρεις φορές, πρέπει να προσαρμοστεί σε έξι διαφορετικά συστήματα ασφάλειας. Αυτό οδηγεί σε καψονάρισμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι δεν τα βλέπουμε απ' έξω αυτά δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. Αντίθετα, θέλουμε να διαμορφωθεί πιο αποτελεσματικά η λειτουργία τους, λιγότεροι κανόνες από όλους αυτούς που υπάρχουν σε όλα αυτά τα κράτη και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να αυξηθεί η αποδοτικότητα, η οικονομική αποδοτικότητα των σιδηροδρόμων. Αυτό σημαίνει ότι έτσι θα αυξηθεί και η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Δεύτερον, να λάβουμε υπόψη το θέμα του περιβάλλοντος διότι η έλλειψη λειτουργικότητας των, των σιδηροδρόμων ευνοεί άλλα μέσα μεταφοράς, άλλες μορφές μεταφοράς που είναι πολύ λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Ξέρετε ότι ε, εάν αναγκάζουμε, όπως είπαμε, ότι αν αναγκάζουμε σε αυτούς που πηγαίνουν από το Βέλιο στο Λουξεμβούργο, τους αναγκάζουμε επί έξι μήνες ε, να κατεβαίνουν από το τρένο στο ε, Αρλόν και να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, τελικά θα παίρνουν το αυτοκίνητό τους απλά και μόνο. Αυτό ε, πρέπει να το καταλάβουμε και γι' αυτό τον λόγο από το Λουξεμβούργο στις Βρυξέλλες θέλουμε τον ίδιο χρόνο εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο δεν αυξάνεται η αποτελεσματικότητα τόσο δεν θα δημιουργούμε και θέσεις απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε στόχους και να μην ε, είμαστε πάντα βυθισμένοι στα τεχνολογικά θέματα. Ως βουλευτές ξέρουμε ότι μπορεί να έρθει ένας ε, εμπειρογνώμων και να μας πει το τάδε είναι τεχνικός εφικτό και ο άλλος, μετά από δύο λεπτά, ο άλλος εμπειρογνώμων να μας πει δεν γίνεται. Θα πρέπει να δώσουμε καθήκοντα στους ειδήμονες, αλλά όχι να κάνουμε τη δουλειά τους. Τελευταίο, Ε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να ε, ασχολούμεθα για μήνες με μια τεχνολογική λύση και μετά να μας λένε δεν είναι επαρκώς ασφαλής. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει σαφής πλειοψηφία και ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε και έναν του κοινού το τέταρτο πακέτο αυτό. Αγιάλα Σέντερ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση αυτή για τη διαλειτουργικότητα έτσι όπως την, την υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το αναγκαίο για να ξεπεραστούν τα ιστορικά εμπόδια που υπάρχουν και γι' αυτό υπάρχει στην τέταρτη δέσμη μέτρων η διαλειτουργικότητα. Σε αυτή τη δέσμη όμως έχουμε το τεχνολογικό πυλώνο και έχουμε προχωρήσει εκεί διότι ε, τα της αγοράς ε, και τα της διακυβέρνησης θα ήταν πιο περίπλοκα. Όμως με απελπίζει το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις συσκέψεις και τις συνεδριάσεις δεν πάμε στα της διαχείρισης και της διακυβέρνησης, γιατί ήδη ως προς τη διαλειτουργικότητα προβάλλονται πτυγές ισχυρού προστατευτισμού, υψώνονται εμπόδια, υποτίθεται με την ασφαλιστική δικλίδα ότι είναι πολύ ιδιαίτερος αυτός ο κλάδος και θα πρέπει υποτίθεται να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Ναι, αλλά είναι η τέταρτη δέσμη που προτείνεται και χωρίς να έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα. Πάντοτε όλη αυτή η επιχειρηματολογία ε, δεν οδηγεί πουθενά, όπως και στην πρώτη δέσμη. Στο τελευταίο φόρουμ που είχαμε υπήρχαν διάφοροι που ε, παρουσίαζαν παράπονα έχουμε ευρωπαϊκούς, κανόνες αλλά δεν έρονται οι εθνικοί κανόνες οι οποίοι προστατεύουν τις εθνικές αγορές. Ό,τι και να προσπαθείτε εσείς να κάνετε άνωθεν ε, δεν αλλάζουν τα πράγματα στη βάση. Βέβαια εγώ είμαι εκφύσεως αισιόδοξη και πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε, να σηκώσουμε τα μανίκια και να καταφέρουμε να άρουμε τους εθνικούς ε, φραγμούς ή περιορισμούς. Συνεχώς μας λένε ότι οι προθεσμίες είναι εξαιρετικά σύντομες, ότι οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν και μάλιστα πολύ ενεργά. Εγώ θα ήθελα να πω στις, στους εθνικούς φορείς το εξής. Αν θέλετε να καταργήσουμε τον ενίο συνδυοδρομικό χώρο και να είστε εσείς οι εθνικοί φορείς ε, αρμόδιοι για την πιστοποίηση μονοπευθυντική θηρίδα, δηλαδή όπως τα τελωνία. Να μπει όποιος ενδιαφέρεται από ένα εθνικό σημείο και εκεί να πιστοποιείται και αυτή η πιστοποίηση να ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Και αυτό θα ήταν μια πρόταση. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Μπιλμπάου ότι δηλαδή πρέπει να ε, ομονοήσουμε και να συμφωνήσουμε ως προς την εκτίμηση της κατάστασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια προσπάθεια, προσπαθεί να ξεπεράσει ε, τους εθνικούς περιορισμούς και φραγμούς. Οι πρώτες αντιδράσεις όμως σε αυτό είναι αντιδράσεις ε, που προβάλλουν πολλές επιφυλάξεις και αυξημένο επίπεδο εθνικής προστασίας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν σημαντικό και το τροχαίο υλικό θα μπορούσε να συμβάλλει στην διαλειτουργικότητα. διότι λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι πέρα από τα εθνικά σύνορα και τα εσωτερικά σύνορα έχουμε δύο μεγάλες ζώνες στον ενίο σιδηροδρομικό χώρο. Μια μεγάλη περιοχή όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε και να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τροχαίο υλικό και μια άλλη ε, περιοχή όπου οι φορείς εκμετάλλευσης ε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα ήθελαν γιατί οι διαχειριστές των υποδομών δεν έχουν το κατάλληλο τροχαίο υλικό που θα επέτρεπε όλες αυτές τις αλλαγές και τη διασύνδεση μεταξύ των δύο αυτών ζωνών και περιοχών. Θέλω να συνεργαστώ όσο θα το περισσότερο και με την κυρία Πελιμπάο και με τους λοιπούς, αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί δεν μας ενθαρρύνουν ιδιαίτερως. Ευχαριστώ κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ την κυρία Μπιλμπάου και θα συνεργαστούμε καλά οι συγητές και οι συγητές, αλλά δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Βεβαίως και ευχαρίστως θα υπάρξει αυτή η συνεργασία. Συμφωνούμε για το στόχο. Θέλουμε ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Γιατί η κατάσταση όπως είναι τώρα, ε, ξέρετε ότι οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί σε όλες τις χώρες είναι οι τελευταίοι εθνικιστικοί οργανισμοί. Εάν δεν τα καταφέρουν, θα εξαλειφθούν. Το μέλλον των σιδηροδρόμων είναι ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε διαλειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και θα πρέπει να μειώσουμε και το κόστος. Μόνο τότε έχει μέλλον ο σιδηρόδρομος. Το status quo δεν μπορεί να διατηρηθεί. Το καταλαβαίνουν όλοι και οι Κομισιόν ακόμη και οι οργανισμοί σιδηροδρόμων ε, το παραδέχονται, αλλά όταν τους ζητάμε να αλλάξουν ε, είναι λίγο πιο δυσκίνητοι. Έχουμε την... Ε, έχουμε την πολλαπλή συμμόρφωση. να σας δώσω παραδείγματα. Λέμε ότι σε όλους τους σταθμούς θα πρέπει ε, να κατεβαίνουν από τα τρένα οι άνθρωποι χωρίς να χρειαστεί να ανέβουν ή να κατέβουν, είναι στο ίδιο επίπεδο δηλαδή. Αλλά δυστυχώς στο νέο σιωδομικό σταθμό στην ε, Στουτγάρδη όντως θα υπάρχει διαφορά επίπεδο ανάμεσα στην, ε, στο επίπεδο του ε, των τρένων και των ε, αποβαθρών. Και έχουμε πει επίσης ότι ε, γίνονται και νέα τμήματα σιδηροδρόμων συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση που δεν είναι παρκός ε, διαλειτουργικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η πρόταση είναι η διαλειτουργικότητα ε, να είναι η διαλειτουργικότητα να είναι αρμοδιότητα του αέρα. Και φυσικά η ΕΡΑ το, δεν μπορεί να αναλάβει όλα τα καθήκοντα των εθνικών οργανισμών. Το θέμα είναι τι θα γίνει σε περιπτώσεις ε, διαφωνιών. Οι εθνικοί οργανισμοί ξέρουν βεβαίως ότι θα υπάρχει ένας ε, επικείμενος οργανισμός από πάνω τους, δεν θα μπορούν λοιπόν να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχουν και προβλήματα βεβαίως ασφάλειας γι' αυτό, αλλά και διαλειτουργικότητας. Αλλά ο αυτός ο επιπλέον οργανισμός, ο από πάνω, θα έχει την ε, τελευταία λέξη σε περίπτωση διαφωνιών. Το TSI που αναφέρθηκε, αυτά τα TSI πρέπει να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι εξαιρέσεις. Στόχος μας πρέπει να είναι λοιπόν αυτός. Και τελευταίο σημείο ε, για τα θέματα που αφορούν την διαλειτουργικότητα. Παίζει ένα ρόλο και το επίπεδο του θορύβου και των ε, ρήπων. Είναι σημαντικός ο ρόλος ε, αυτός γιατί και αυτός προκαλεί στερευλώσεις του ανταγωνισμού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ρήπων. Πρέπει να υπάρξουν οριακές τιμές. Γιατί αν δεν μειώσουμε τις εκπομπές και για το θόρυβο και για τους ρήπους ε, και πρέπει να οδεύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων έχει είναι σαν στόχο να συζητήσουμε τις τεχνικές πτυχές ε, της πρότασης ε, της Κομισιόν. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων, να δούμε πού θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα, ποιες λύσεις ε, θα μπορούσαν να βρεθούν, τι δυνατότητες βελτίωσης της πρότασης της Κομισιόν υπάρχουν για την διαλειτουργικότητα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σε επίπεδο συμβουλίου το project αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Αντίθετα βέβαια με τον κανονισμό για την ασφάλεια και για την ε, Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, το ΕΡΑ. Όμως πιστεύω ότι ε, για την ανάπτυξη του τεχνικού τομέα έχει επιτευχθεί πρόοδος. Για την διαλειτουργικότητα το βασικότερο πρόβλημα συνδέεται με τις διαδικασίες και τις ευθύνες. Ποιος είναι υπεύθυνο γιατί και ο ΕΡΑ δεν μπορεί να αναλάβει όλες τις ευθύνες. Αυτός ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση πρέπει να είναι και ο υπεύθυνος, κυρίως εάν και εφόσον μια κάποια απόφαση είναι λανθασμένη. Διότι αλλιώς δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι κατανοητές, διάφανες και δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα σταματήσουν να υπάρχουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσο θα περιορίσουν την προσβασιμότητά του στην αγορά οι εθνικοί οργανισμοί. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Παγνιό για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συμμερίζομαι την ανάλυση της Κομισιόν όσον αφορά την βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος για την αδειοδότηση, όμως για την οδηγία για την διαδηλειτουργικότητα οι προτάσεις δεν είναι σωστές, δεν είναι κατάλληλες, διότι αντί να αυξήσουμε τη συμβατότητα, αν θέλετε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και τις εθνικούς οργανισμούς, ε, αυξάνουμε τις δυσκολίες ε, και τις υποχρεώσεις. Ε, θα πρέπει ο ΕΡΑ να παίξει έναν ρόλο μοναδικού συνομιλητή αν θέλετε με τους ε, εθνικούς οργανισμούς και να παίξει και τον ρόλο χωροφύλακα. Η, η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα μπορούσε να γίνει το, η μοναδική πύλη αν θέλετε για να ε, ελέγχει τα, τα οχήματα τα οποία θα περάσουν τουλάχιστον κάποιο ευρωπαϊκό σύνορο. Από εκεί και πέρα οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να αξιολογηθούν με βάση τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης. Ε, εάν γίνει η τροποποίηση αυτής ε, της ε, οδηγίας θα πρέπει ε, πρόεδρε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χορηγούνται οι άδειε για τα, υποσυστήματα και τα οχήματα. Η ανησυχία μου έγκυται στο γεγονός ότι σε περίπτωση παράδοσης η αδειοδότηση για την κυκλοφορία στην αργορά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και δεν γίνονται οι δοκιμές για να ελεγχθεί η τεχνική συμβατότητα ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο υλικό. Επίσης ανησυχώ διότι δεν συνδέεται πλέον ο έλεγχος με τον εξοπλισμό ή το μηχάνημα αλλά με την εταιρεία κατασκευής. Επίσης δεν αναφέρονται και οι συνθήκες κατά τις οποίες η άδεια μπορεί να αφαιρεθεί ή να περιοριστεί. Και αυτό με ανησυχεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πολλούς ε, Α, ο κύριος Σπάκ, γιατί υπάρχουν πολλοί ομιλητές για την διαλειτουργικότητα. Αν θε, επίσης να σηκώνετε και το χέρι σας, διότι δεν διαβάζω το, μυαλό σας ε, ούτως ή άλλως. Ο κύριος Σπάκ, και δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όπως άκουσα και όπως ξέρω υποστηρίζουμε όλοι τις προσπάθειες ε, για να βελτιωθεί η ασφάλεια στους σιδηροδρόμους να μην κάνουμε το λάθος επειδή δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνιστικότητα να μειώσουμε την ε, ανάγκη ασφάλειας. Η ασφάλεια βασίζεται στις εθνικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν ε, τη λειτουργία των σειροδρόμων αλλά και τους τεχνικούς κανόνες και εδώ περιμένω και από τον κλάδο συνέπεια. Ξέρετε ότι γίνεται προσπάθειες να προστατευτούν κάποια συστήματα. Ε, δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Η ασφάλεια τι σημαίνει. Να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα, να βελτιωθεί αυτός ο οργανισμός ιδιοδρόμων και να υπάρξει οδηγία για την ασφάλεια. Οι διάφοροι φορείς πρέπει να καθορίσουν σαφώς ρόλο και ευθύνες. Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από ε, ασάφεια για το ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Δεν υπάρχει ακόμη ε, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς και δεσμευτικοί κανόνες για τη συντήρηση, την πιστοποίηση κτλ. Και επίσης οι κοινωνικές συνθήκες ε, είναι πολύ επιφανική η πρόταση της Κομισιόν στον τομέα αυτό. Δεν ε, καθορίζονται τα, οι αρμοδιότητες, η κατάρτιση. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Περνάμε στο επόμενο σημείο για την ασφάλεια. Ε, δεν έχουμε άλλη διαλειτουργικότητα. Ο Μάικλ για έξι λεπτά. Λοιπόν, η ασφάλεια παίζει μεγάλο ρόλο. Και ε, γενικώ βεβαίω δεν θέλουμε να μειωθεί η ασφάλεια. Θέλουμε το μέγιστο ε, επίπεδο ασφάλειας. Ωστόσο, ωστόσο, εάν οι άλλες μορφές ε, μεταφορών ήταν τόσο ασφαλείς όπως είναι τώρα ο σιδηρόδρομος, τότε θα ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση. 40.000 άτομα πεθαίνουν στους δρόμους κάθε χρόνο. Αλλά για τους σιδηροδρόμους, εάν γίνει ένα ατύχημα, γίνεται τρομερή παρουσίασή του από τον τύπο. Αυτό είναι καλό. Αλλά να μην αγνοούμε και τις άλλες μορφές. Εδώ υπάρχει δυσαναλογία, τονίζω. Οι σιδηρόδρομοι είναι ασφαλές μέσω μεταφοράς. Αυτά τα πιστοποιητικά που προτείνει η Κομισιόν για την ασφάλεια περιέχουν ότι οι οργανισμοί σιδηροδρόμων θα πρέπει να είναι κύριοι των διαδικασιών. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν να ελέγξουν, να έχουν το αναγκαίο υλικό, το αναγκαίο προσωπικό κτλ. Τι λείπει όμως, η απόδειξη της ασφάλειας. Βεβαίω έχω αυτό το πιστοποιητικό ω επιχείρηση, αλλά αν λειτουργεί σωστά αυτό το οποίο δημιούργησα, εάν είναι αρκετά καλά τα άτομα, καταρτισμένα, εδώ πρέπει να γίνουν περισσότερα. Εδώ λέμε αν υπάρχει σχέδιο για το πως πρέπει να γίνουν όλα αυτά, θαυμάσια. Όχι. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο σχέδιο και διαδικασίες Θέλουμε να έχουμε την εγγύηση ότι όντως και τα άτομα κατέχουν τις διαδικασίες αυτές Δεύτερον, τα πιστοποιητικά ισχύουν σε όλη την Ένωση. Αυτό το έχουμε πει και για την ε, διαποδοχή. Δηλαδή, εάν μια, ε, ένας είναι καλός, ε, θα πρέπει να είναι καλός παντού και αν σε κάποια χώρα δεν ε, θεωρείται καλός, θα πρέπει να αιτιολογείται. Έτσι νομίζω ότι κερδίζουμε χρόνο. Θέλουμε λοιπόν να ισχύσει σε όλη την ε, Ένωση. Αλλά κάποιοι λένε όχι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο και η Γερμανία και η Γαλλία εάν συμφωνούν ε, εντάξει να έχουν ένα επίπεδο η Πολωνία, η Τσεχία και η Σλοβακία ένα άλλο, οι Βαλτικές χώρες άλλο. Όχι, να μην χάσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Θα πρέπει να ισχύουν αυτές οι πιστοποίησεις για όλη την Ένωση. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν εθνικές ιδιομορφίες. Σαφές. Δεν μπορούμε να τα ρυθμίζουμε όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά σε περίπτωση διχογνωμιών την τελευταία λέξη πρέπει να το έχει το αέρα. Να ξέρουν οι εθνικές αρχές ότι δεν έχουν την τελευταία λέξη. Γιατί η αέρα πρέπει να έχει και την τελική ευθύνη. Έχει δίκιο ο κύριο Μπαχ. Αν ε, είναι μοιρασμένη η ευθύνη δεν υπάρχει. Η αέρα πρέπει να αναλάβει σε περιπτώσεις διχογνωμιών την τελική ευθύνη. Αλλά θα πρέπει να ακούσει τις εθνικές αρχές, να πει ε, γιατί έχετε αντιρρήσεις, να μην πει ότι αν υπάρχουν άλλα χρώματα για κάποια φανάρια αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Τώρα η τάση του ρεύματος. Βεβαίως, ε, πρέπει να έχει περισσότερη ε, πρόσβαση στην αγορά. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μειώνει την ασφάλεια. Πρέπει να είναι σαφές. Ξέρω ότι ο Γερμανικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων στις αναλύσεις τους επιδιώκει 100% ασφαλείας. Αν το έκαναν αυτό ε, στους δρόμους δεν θα μπορούσε να κινηθεί κανένα αυτοκίνητο. 100% ασφάλεια ε, στις οδικές μεταφορές δεν ισχύει. Ούτε και στους σιδηροδρόμους παρά το ότι γίνονται πολύ, συμβαίνουν πολύ λιγότερα ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ανάλυση των κινδύνων, να αποφύγουμε τους κύριους κινδύνους. Αλλά αν θέλουμε 100% ασφάλεια, τότε δεν θα πρέπει να βγω από την αίθουσα, γιατί μπορεί να μου πέσει κάτι στο κεφάλι βγαίνοντα. 100% ασφάλεια δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά θέλουμε την υψηλότερη εφικτή ασφάλεια. Δεν πρέπει να μειωθεί σίγουρα η ασφάλεια. Βεβαίως ευρωπαϊκοί κανόνε δεν πρέπει να βασίζονται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αντίθετα, θέλουμε να αυξηθεί η ασφάλεια. Παρά το ότι οι σιδηρόδρομοι έχουν υψηλό ποσοστό ασφάλεια. Με αυτέ τι ε, κατευθύνσει θα διατυπώσω την έκθεσή μου. Επί τη αρχή νομίζω συμφωνούμε και προσβλέπω και στι ε, παρεμβάσει σα. Από ότι ξέρω τη συνεργασία μα νομίζω ότι θα επιτύχουμε μια καλή έκθεση, θα επιτύχουμε συμβασμού για να προωθήσουμε τους σιδηροδρόμους, θέλουμε να αυξηθεί η κινητικότητα του πληθυσμού, να προστατεύσουμε και το περιβάλλον, όλα αυτά επιτυγχάνονται μόσο ενίσχυση των σιδηροδρόμων. Εάν οι σιδηρόδρομοι αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχή τους μεταφορές, επειδή οι σιδηρόδρομοι έχουν τεράστιο κόστος για τις ε, σταθερές εγκαταστάσεις, εάν αυξηθούν λοιπόν το ποσοστό επιβατών και ε, αγαθών που ε, μετακινούνται μέσω ε, σιδηροδρόμου θα έχουμε και μεγάλες εξοικονομήσεις όπως βλέπουμε στις ΗΠΑ διότι επειδή είναι ακριβώς το κόστος των εγκαταστάσεων όσο λιγότεροι μετακινούνται ε, μέσω σιδηροδρόμων τόσο υψηλότερο είναι το κόστος αναμονάδα. Ε, στον τομέα αυτό επειδή εμεί έχουμε μόνο 17% μέσω σιδηροδρόμων και οι ΗΠΑ 40%, οι ΗΠΑ αποτελούν υπόδειγμα. Ίσως άλλο το μισό, όχι σε αυτόν ναι. Ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά ο George. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για αυτό τον συντροματικό χρόνο. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη είπα. Ένα-δύο θέματα. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αίρα και εθνικών οργανισμών είναι πολύ σημαντικό να καθοριστεί σαφώς να καθοριστούν τα όρια βεβαίως ε, το αέρα ούτε μπορεί ούτε θα πρέπει να τα ρυθμίζει όλα στο μέλλον και στο μέλλον οι εθνικές αρχές ασφαλείας θα έχουν πολύ σημαντικά καθήκοντα. Ο Μάικλ μίλησε για τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, TSI. Βεβαίως πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε για αυτά. Μιλάμε για τις 11-12 χιλιάδες ρυθμίσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εάν όμως αυτά τα TSI γίνουν πραγματικότητα, και αν ε, συνδυάζονται, γίνει εφικτό να συνδυάζονται οι εθνικές προδιαγραφές με αυτά τα TSI, τότε θα μειωθούν οι εθνικές ρυθμίσεις. Για τα τεχνικά συστήματα και το τροχαίο υλικό και τις υποδομές ε, πρέπει να υπάρξουν ε, πιο μακροπρόθεσμες προθεσμίες, ούτως ώστε για το νέο υλικό που θα αγοραστεί, αλλά και για το υπάρχον υλικό, να μην υπάρξει τρομερά μεγάλο κόστος. Δεν πρέπει να απαιτήσουμε όλα να αντικατασταθούν πολύ βραχυπρόθεσμα. Είπα λοιπόν, πρέπει να καθοριστεί σαφώς ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Κάτι που ανέφερε και ο κύριος Γκρός, για να καταλάβουμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα που δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν τα προβλήματα μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου. Οι Λουξεμβούργοι για τις πιο ακραίες περιπτώσεις έχουν πέντε διαφορετικά ε, ε, συστήματα ασφαλείας ε, στους ιδιοδρόμους τους, τους κινητήρες, ενώ το Λουξεμβούργο έχει επενδύσει μαζί με την Δανία και την Ελβετία, έχει επενδύσει για ένα επαρκές και πολύ προηγμένο σύστημα ασφαλείας, το οποίο όμως δεν δέχονται οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Βέλγοι. Βεβαίως, οι Βέλγοι πριν από έξι μήνες ε, ζήτησαν ε, να γίνουν νέοι έλεγχοι ασφαλείας, πρέπει να κάνουμε νέα τεστ, ε, πρέπει να υποβάλουμε τις έγκρισεις, πρέπει να το ανακοινώσουμε, να το κοινοποιήσουμε στους Βέλγους και μάλιστα δεν ξέρουμε σε ποιον πρέπει να το ανακοινώσουμε στους Βέλγους, να το κοινοποιήσουμε. Είναι η ή SNCB αρμόδιοι. Και περιμένουμε να τα κάνουμε εμείς όλα αυτά. Πρέπει αυτούς, αυτές τις διαδικασίες να τις σταματήσουμε επιτέλους. Στο μέλλον πρέπει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες. Εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του οργανισμού αέρα, όπως για παράδειγμα στις αεροπορικές μεταφορές. Λειτουργεί. Θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και στον τομέα των σιδηροδρόμων. Ευχαριστώ πολύ. Αγιάλα Σέντερ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη μελέτησα με ενδιαφέρον ως προς την οδηγία για την ασφάλεια και τις αλλαγές που θέλει η Κομισιόν να επιφέρει. ήταν πλέον καιρός να γίνει κάτι τέτοιο να έχουμε νέο πιστοποιητικό ασφαλείας που να ισχύει σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όταν λέμε κάτι τέτοιο, διάφοροι αντιδρούν και λένε ότι όχι δεν θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο ασφάλειας και βεβαίως εμείς θέλουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Άλλωστε τα τρένα είναι το πιο, και θεωρείται το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Αυτό χρησιμοποιούν οι εθνικοί φορείς εκμετάλλευσης ως άλοθη για να θέσουν νέους φραγμούς, περιορισμούς, ώστε τελικά να μην οριμάσει το σύστημα και να μην φτάσει σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό. Το οποίο βεβαίως θα εξασφάλιζε την πλήρη διαλειτουργικότητα και την πλήρη ασφάλεια. Νομίζω ότι οι δύο οδηγίες πρέπει να έχουν συνοχή μεταξύ τους και θα πρέπει εμείς να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Συμφωνώ με τον κύριο Μπακ. Χρειάζεται η ασφάλεια όχι μόνο στην οδηγία για τη διαλειτουργικότητα, αλλά και η κοινωνική δέσμη μέτρων είναι σημαντική. Δηλαδή να υπάρξει μία δέσμη κοινωνική μέσα σε αυτή την τέταρτη δέσμη για το σιδηρόδρομο ώστε να λέμε ξεκάθαρα ότι θα λυθεί ε, αυτό το τεράστιο δίλημα που πάντοτε προκύπτει με τις αναδιαρθρώσεις. Κάτι το οποίο καθυστερεί τα πράγματα και αποτελεί τροχοπέδι. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των δράσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ασφάλεια και θέλουμε να είναι ενισχυμένη η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Εάν πάμε προς την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφαλείας, τότε είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πεδίο υπευθυνότητα και σε περίπτωση ατυχήματος. Υπό αυτή την έννοια και μαθαίνοντας από τις εξελίξεις που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό, θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αρκετά τη διατύπωση ώστε η ασφάλεια να συνάδει και με τη διαλειτουργικότητα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπένιεν εξ ονόματος των Φιλελεύθερων. Τέσσερα λεπτά. Δεν χρειάζομαι τέσσερα λεπτά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συνένεση είναι αρκετά ευρία εδώ και θα είναι πιο εύκολο ε, να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Κοινοβούλιο παρά αλλού. Όπως είπε και η κυρία Αγιάλα Σέντερ, πράγματι θα υπάρξουν αντιστάσεις. Θα υπάρξουν άλλοθη και δικαιολογίες που θα προβάλλουν οι εθνικοί φορείς οι οποίοι ο καθένας θα λέει ότι το δικό του σύστημα είναι το πιο ασφαλές και ότι οποιαδήποτε εναρμόνιση ε, θα πλήξει την ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να κάνουμε το παν ώστε να αντιστρέψουμε αυτά τα επιχειρήματα που μας εμποδίζουν να προοδεύσουμε. Συμφωνώ με τα σχόλια του Μάικλ για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Νομίζω ότι θα είναι το κλειδί το ευρωπαϊκό ε, πιστοποιητικό. πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο χρήσης των συνδροδρόμων για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το κόστος της χρήσης του. Και θα το πετύχουμε αυτό με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες λαμπρές εξαιρέξεις, όπως είναι το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όμως το βασικό πιστοποιητικό ασφάλειας μπορεί να ισχύει σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια με ειδικέ προδιαγραφές για ειδικά δίκτυα και για κάποια ειδικά συστήματα, επασφελτώσει ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα, να διασφαλίσουμε επίσης ότι μειώνονται τα κόστη, διατηρείται η ασφάλεια, αλλά δεν υπάρχει και γραφειοκρατικό άχθος. Είναι, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός ο σιδηροδρομικός κλάδος στην Ευρώπη. Η διαδικασία επιστοποίησης λέει ότι απαιτείται όλες τις μορφές ανανέωσης ή αναβάθμισης των αδειών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τις ελάσσονες ανανεώσεις και αυτές να μην χρειάζεται για να τις πάρει κανείς εκ νέου επιστοποίηση. Τι σημαίνει ελάσσονα ανανέωση. Αν κάθε ανανέωση πρέπει να υπάγεται σε μια διαδικασία καινούρια πιστοποίησης, ε, νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση που δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεση. και άλλα ζητήματα θα προκύψουν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων ως προς το τροχαίο υλικό, το εφιστάμενο και το επιχείρημα του κυρίου Μπακ. Να μην επιτρέψουμε την εθνική πιστοποίηση σε υπερβολικό βαθμό. Με το υφιστάμενο τροχαίο υλικό Πολλοί από αυτό ίσως δεν μπορεί να ε, πάρει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κόστος συνεπάγεται όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά κυρίως ήθελα να πω ως προς το νέρα και σημαντικό είναι και το θέμα των εθνικών αρχών ασφαλείας και η σχέση τους με ε, τον αέρα. Θα πρέπει να υπάρξει μια κάποια ρύθμιση ή διευθέτηση τύπου υπεργολαβίας, subcontracting. Και ε, αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα ε, για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα έχοντας ταυτόχρονα και τη συγκατάθεση των κρατών μελών. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας μια ομάδα επισκεπτών κατόπιν πρόσκλησης ε, της κυρίας Αγιάλα Σέντερ ε, στην Ισπανία από τις αγροτικές περιοχές της Αραγωνίας. Είναι οι επισκέπτες μας. Καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέροντα τα θέματα που μας απασχολούν στην Επιτροπή μας. Έχω κι εγώ πάει στην Αραγωνία. Είναι μια πανέμορφη περιοχή Είχα αυτή την ευκαιρία να την επισκεφθώ. σα καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη διανομή. Ο κύριος, διαμονή με συγχωρείτε. Ο κύριος Ζήλερ, τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ για σε αυτό το σύστημα, νέο σύστημα πιστοποίησης και την έκθεση του κύριου του πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ε, το, το τμήμα Β, ότι το τμήμα Β του πιστοποιητικού δεν θα πρέπει να δεν θα εξαφανιστεί, το τμήμα Α θα παραμείνει και αυτό θα πρέπει να γίνει ε, σεβαστό από, το, από όλους τους εθνικούς οργανισμούς. Ε, έχετε δει το πρώτο τμήμα. Εγώ το έχω δει και τα, έχω δει και τα δύο. Το πρώτο τμήμα αφορά την άδεια λειτουργία, αν θέλετε, σε κάποιου τομεί. Το Β όμως είναι ένα συνοθήλευμα διαφόρων στοιχείων. Επομένω, εάν θέλουμε τα πάντα να παραπέμψουμε στην αίρα, μήπω θέτουμε σε κίνδυνο τους κανόνε ασφάλεια. έστω και αν το εύρο των συνδρομικών τροχιών είναι το ίδιο παντού, ε, δεν ξέρω, στη Σουηδία τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στην κεντρική Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την ε, ασφάλεια ε, εξαφανίζοντας το, το Β, για το τμήμα Β, διότι το τμήμα Β το, χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιούν συχνά σαν πρόφαση. Αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα και τα πάρα πολύ σημαντικά επίσης. Ο κύριος Φιντάνσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν για την διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και τον ρόλο της ΕΡΑ ε, προχωρεί στη σωστή κατεύθυνση. Κατεύθυνση διαπλούστευσης ε, ε, κεντρικής διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο το, της χρήσης και της θέσης σε λειτουργία του υλικού και του, του εξοπλισμού. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και σε εθνικό επίπεδο ε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες εθνικές ε, διατάξεις ε, που δημιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, περιορίζονται οι προθεσμίες και περιορίζεται και το κόστος χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε, δεν θα πρέπει τα θέματα το, της πιστοποίησης του υλικού, της αδειοδότησης κτλ. να επανέλθουν σε εθνικό στις εθνικές αρχές. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με κάποιο τρόπο έναν, ε, το καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην ΕΡΑ και στους εθνικούς οργανισμούς και οι προθεσμίες να περιοριστούν σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση τουλάχιστον. Τώρα όσον αφορά τις προθεσμίες ε, για την ε, θέση σε λειτουργία στην κοινωτική αγορά θα πρέπει οι προθεσμίες να περιοριστούν εξασφαλίζοντα την ασφάλεια βέβαια και η ΕΡΑ θα πρέπει να έχει το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει να είναι επανδρομένη κατάλληλα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αρμοδιότητες ε, που, τους, ε, που τις έχουμε δώσει. Επίσης η μετάβαση ανάμεσα στο παλιό σύστημα και στο νέο σύστημα θα πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι εθνικές διατάξεις ε, και απαιτήσει θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΕΡΑ. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι ε, θα πρέπει να γίνει μία σαφής αναφορά σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες ε, στο, για τις συνδρομικές μεταφορές και να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι υπεύθυνο, όχι ενδεχόμενα ο κάτοχος του υλικού. Μην ξεχνάτε το ατύχημα την τραγωδία του Διαρέτζο και εκεί είχαμε ένα τέτοιο θέμα ε, ευθύνης. Ποιος έχει την, την ευθύνη για το, για υλικό. Ο ιδιοκτήτης στο οποίο στο κυκλοφορεί. Κύριε Σπαγνιό, για δύο λεπτά, αγαπητέ αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα πω και εγώ τι προσωπικέ μου απόψει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πιστεύω ότι είναι πρόωρο η ΕΡΑ να αντικαταστήσει πλήρως τις εθνικές αρχές αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα πρότεινα να υπάρξει ένα σύστημα όπου θα υπάρχει ένα σύστημα ε, υποβολή εφέσεων αν θέλετε σε περίπτωση που υπάρχουν και στο εθνικό σύστημα και ο ρόλος των εθνικών αρχών δεν μπορεί να περιορίζεται απλώς και μόνο σε μία αποστολή ε, προαιρετικής ε, ε, προαιρετικού ελέγχου και εξπόστο για ε, ελέγχου των αδειών που ε, χορηγεί η ΕΡΑ. Θα πρέπει οι εθνικές αρχές να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ε, αρχιτεκτονική ελέγχου της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας έτσι ώστε να εφαρμόζονται σωστά οι εθνικοί κανόνες αλλά και να υπάρχει ένα ορισμένο σύστημα για την χορήγηση των πιστοποιητικών και των αδειών. Ευχαριστώ. Αυτά... Α, εάν έχουμε χρόνο θα δώσω το λόγο ξανά στους ε, εισηγητές. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, είναι διαδικαστικό ή όχι. Όχι για την αίρα ήθελα να πω κάτι. Πρόεδρος, θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή και μετά θα μιλήσουν τα μέλη για την αίρα. Λοιπόν, για την αίρα, Ρόμπερτς, 6 λεπτά. Όλοι θέλουν να δημιουργηθεί αυτό το, αυτή η αίρα Επομένως, σε ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και χαίρομαι που οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό το θέμα, τρίτος πυλώνος αν θέλετε, είναι μία σύνοψη των προηγουμένων ε, θεμάτων που μας απασχόλησε, διαλειτουργικότητα και ασφάλεια. Επομένως ε, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο πιστεύω να καταλήξουμε σε μία συμβαστική πρόταση για τον τρόπο και για το λειτουργία και για το εύρος ε, των αρμοδιοτήτων του, της ΕΡΑ αποκτά και κάποιες νέες ε, αρμοδιότητες, παραδείγματος χάρη την ε, χορήγηση ε, του εννοέου πιστοποιητικού για τους φορείς που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης για την πιστοποίηση του εξοπλισμού του τροχαίου υλικού, των σημάτων των ενδείξεων ενδείξεων που βελτιώνουν το όλο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ε, εάν χρειαζόμαστε μια κάποια μεταβατική περίοδο για τις νέες αρμοδιότητες που αποκτά η ΕΡΑ. Η Κομισιό αυτή τη στιγμή δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο. Όμως ε, βλέπουμε την ισχύ στις αεροπορικές μεταφορές και εκεί υπήρχε ε, στην αεροπορία υπήρχε μεταβατική περίοδος και συλλειτουργούσαν για κάποια περίοδο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία και οι Εθνικές Υπηρεσίες. Δεν θα εξαφανιστούν ε, βέβαια οι Εθνικές Υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες δεν έχουν ε, εκχωρηθεί ακόμα στην αίρα Επίσης, ποιος πληρώνει τι. Υπάρχουν χώρες όπου τα πιστοποιητικά χορηγούνται δωρεάν και χρηματοδοτούνται από τον Εθνικό Πρωτολογισμό, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Εμείς έχουμε σαν καθήκον να βρούμε μια λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον πελάτη. Ο πελάτης ε, μπορεί να είναι ή ο κατασκευαστής ή η συνδρομική εταιρεία. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις. Ή το πιστοποιητικό να χορηγείται από την ΕΡΑ με κάποιο τίμημα και το πιστοποιητικό αυτό θα ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ή η δεύτερη εναλλακτική λύση θα είναι εάν η συνδρομική εταιρεία δεν είναι τόσο φιλόδεξη και θέλει να περιοριστεί μόνο στο, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, θα μπορεί να έχει την δυνατότητα να παίρνει το πιστοποιητικό από τον εθνικό φορέα. Εάν δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει επιλογή για τον πελάτη, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει η να οριοθετήσουμε μάλλον τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΕΡΑ από τη μια πλευρά και ο Εθνικός Φορέας από την άλλη. Θα πρέπει και η ΙΕΡΑ να έχει έναν τρόπο συνεργασίας, μια μέθοδο συνεργασίας με, τις εθνικές, με τους εθνικούς οργανισμούς, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, συμπληρωματικά κόστη αλλά και καθυστερήσεις. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου σαν πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες που είμαστε και να βρούμε την κατάλληλη λύση. Μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίος φορέας ενδεχόμενα, ε, αλλά και να δίνεται η δυνατότητα ε, εάν κάποιος ε, θέλει να περιοριστεί μόνο σε μία αγορά, να μπορεί να το κάνει. Εγώ το έχω συζητήσει όχι μόνο με το θέμα με τους συναδέλφους από τις γειτονικέ χώρες της Βαλτικής, αλλά και με την Φιλανδία. Αυτό το εύρος των ε, τροχιών ε, που είναι διαφορετικό, εμφανίζεται και στην Σοβιετική Ένωση. Όμως εκείνες οι αγορές είναι τελείως απομονωμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα πράγματα είναι, η κατάσταση είναι λίγο κατακαιρματισμένη. Το 15-24 επί 24 24 υπαρχει στη Μόσχα αυτή τη στιγμή για το τροχαίο υλικό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει εάν όλα τα καθήκοντα τα αναλάμβανε η ΕΡΑ και δεν θα μπορούσε να πιστοποιήσει αυτό το τροχαίο υλικό, διότι η απόφαση λαμβάνεται στη Μόσχα, παραδείγματος χάρη. Επίσης υπάρχουν και τεχνικά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κάπως ασυνήθιστη κατάσταση, παράλογη κατάσταση όπου στην Λετωνία και στη Λιθουανία ας πούμε οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να ε, περάσουν τα σύνορα ή οι φιλανδικοί σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να πάνε στην Ρωσία. Ελπίζω ότι θα ε, καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζήλερ. Πριν δώσω λόγο στον κύριο Ρικέ να καλωσορίσουμε τους, συναδέλ, συμπατριώτες του κ. Ρικέ που είναι εδώ, που μας επισκέπτονται. Είναι ε, στρατιωτική σε αποστρατεία ε, από μια πόλη που είναι κοντά στο Μέτσα. Ε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας Μεταφορών και Τουρισμού. Ελπίζω να περάσετε καλά στις Βρυξέλλες και να ε, βρείτε να κρίνετε ε, τα όσα διαδραματίζονται εδώ σε αυτή την αίθουσα ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής ε, είναι συμπατριώτης σας, είναι Γάλλος, είναι ο κύριος Ρικέ. Τέσσερα λεπτά κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προηγούμενες παρεμβάσεις για την διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια ε, τα σχόλια του εισηγητή για τον φορέα αυτό, τον οργανισμό αυτό. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε. Όλοι είμαστε υπέρ του σιδηρόδρομου. Όλοι θέλουμε μεγαλύτερη ενοποίηση και περισσότερη ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, εκτός από όταν γίνεται λόγος για το κόστος για τη μεταγραφή αυτή, αυτών των οδηγιών. Εκεί εντοπίζονται οι διαφορές. Ως προς το θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, το οποίο είναι και ο βραχίωνας που συνδέει τη διαλειτουργικότητα με την ε, ασφάλεια και την ποιότητα, το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς από τους κανόνες θα πάμε στο επιχειρησιακό σκέλος. Πού ακριβώς θα τοποθετήσουμε τον ορισμό των κανονιστικών διατάξεων και πώς θα τα μεταγράψουμε αυτά στο επιχειρησιακό σκέλος και στην καθημερινή λειτουργία. Μεγάλη είναι η συμφωνία στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το θέμα των τεχνικών προδιαγραφών ε, διαλειτουργικότητας, των στόχων της ασφάλειας, όλα αυτά μπορούν και πρέπει να καθοριστούν από τον ΕΡΑ. Είναι γενικότερη η συμφωνία ως προς αυτό πιστεύω. Όμως, μόλις άπαξ και γίνεται λόγος για τα εκτελεστικά καθήκοντα, εκεί η συμφωνία δεν είναι τόσο ομόφωνη. Στα πιστοποιητικά ασφάλειας ε, υπάρχει διαφωνία απόψεων ποιος θα εκδίδει τι και σε ποιο επίπεδο. Ο Ρόμπερτ μας ανέφερε τη δική του άποψη ότι πρέπει αυτά να εκδίδονται σε δύο επίπεδο. Μετά για τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις ε, εισόδου στην αγορά υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες. Ο καθένας θέλει να εισαγάγει κάτι για να ε, παρεμποδίσει ή να επιβραδύνει ε, την ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λέγοντας ότι η διαλειτουργικότητα δημιουργεί ταχύτεχνικα προβλήματα ή για λόγους ασφαλείας υπάρχουν τα ψή θέματα, προκειμένου να μην προχωρούμε. Νομίζω λοιπόν ότι Υπάρχει απάντηση σε αυτές τις τεχνικές αντιρρήσεις και βρίσκεται στην οδηγία η οποία θα καθορίζει διάφορα στοιχεία. Πρώτον τα μέσα που θα έχει ο αέρας στη διάθεσή του. Με κάθε ειλικρίνεια σας λέω ότι μελέτησα πολύ προσεκτικά τα παραρτήματα στο κείμενο της Επιτροπής και θεωρώ ότι οι προβολές και οι προβλέψεις της δεν έρονται στο ύψος των περιστάσεων που αρμόζει και ρωτώ για αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει στην εξίσωση να ε, μπουν ε, από τη μία πλευρά τα μέσα που θα έχει ο αέρα και από την άλλη οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει. αλλιώ ε, συνεχώς θα προβάλλονται επιχειρήματα και δικαίως ότι ο αέρα δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, στην ε, διαβίβαση όλων αυτών από τους εθνικούς φορείς στον ΕΡΑ θα πρέπει να συζητηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, το υπονόησαν και οι ορισμένοι συνάδελφοι προηγουμένως, να δώσουμε ένα χρονικό ε, περιθώριο. Οι προσταγές ασφαλείας μας κάνουν ε, να είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέψουμε μια μεταβατική περίοδο. Είναι δύσκολο να το αποφύγουμε αυτό. Και πού θα πρέπει σε ποιο σημείο θα πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των εθνικών φορέων και του ΕΡΑ. Ε, δεν θα εξαφανιστούν οι εθνικοί φορείς, ούτε θα πρέπει να επομιστούν το ρόλο του ΕΡΑ. όσο περισσότερες αρμοδιότητες ανατίθενται στους εθνικούς φορείς, τόσο περισσότερο θα καθυστερεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυτού του κολάδου το σωστό είναι να βρούμε ένα σωστό σημείο ισορροπίας που θα μοιράζονται τα καθήκοντα ανάμεσα στους δύο. Ο πρόεδρος. Έχουμε γαλλική ομάδα, Γάλλους επισκέπτες και ο επόμενος ομιλητής θα είναι Γάλλος από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Παχνιού. Ναι, ε, γαλλική ομάδα. Σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Για να δούμε όμως οι νομοθετικές προτάσεις για το τεχνικό σκέλος είναι απαραίτητες, είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο αυτό. Την αναθεώρηση αυτή την περιμένει το σύνολο του κλάδου εδώ και καιρό. Σήμερα ο κλάδος υποφέρει διότι είναι τεράστια η καθυστέρηση για την έγκριση του τροχαίου υλικού μέχρι και δύο χρόνια και πολύ υψηλό το κόστος αυτού. Συμφωνώ πολύ με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τις βασικές αδυναμίες και τα όρια ε, του ευρωπαϊκού πλαισίου. Και γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του ΕΡΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Σιδηροδρόμων, ο οποίος έχει την έδρα του στη Βαλενσιέν, μια πολύ όμορφη πόλη, και ο οποίος έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη διαλειτουργικότητα και την ε, <clears throat> προστασία ε, της ασφάλειας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες ε, του ΑΕΡΑ για να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αποκλίσεις μεταξύ των 27 εθνικών φορέων. Να χαιρετήσουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν ώστε ο, ΕΟΣ, ο αέρα να είναι η μόνη πύλη ε, για την έκδοση των προστοποιητικών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες, τα μέσα που θα έχει, τα χρηματοδοτικά, αλλά και οι ανθρώπινοι πόροι πάνω στους οποίους θα βασίζεται. Συμφωνούμε με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταργηθούν οι κανονιστικές διατάξεις που πλεονάζουν ή που αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εν τούτης, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να προβλέψει μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα αυξηθούν οι αρμοδιότητες του ΕΡΑ. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο ο ΕΡΑ θα αποκτήσει τους απαραίτητους πόρους και την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη που του που ε, είναι εκ των για να μπορέσει να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να έχει δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε έναν τομέα που έχει άμεσο αντίκτυπα στην ασφάλεια στις υδροδρομικές μεταφορές. Θα πρέπει σιγά σιγά να αναλαμβάνει και σταδιακά προοδευτικά να αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες. Θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε ζητούμε από τη μεταβατική περίοδο για τη σύσταση και οργάνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στις εναέριες μεταφορές. Είχε προβλεφθεί εκεί μεταβατική περίοδος 3,5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέχιζαν τα κράτη-μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά για τα αεροσκάφη. Ε, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο ασφάλειας και να μην υπάρχει διάκριση ε, στις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. Μπορούμε λοιπόν να εμπνευστούμε από το παράδειγμα των εναέριων μεταφορών, ούτω ώστε να έχουμε μια μεταβατική περίοδο, ε, ώστε ε, ο αέρα να αποκτά όλο και περισσότερες αρμοδιότητες κατά τη διάρκεια αυτής. Αυτά έχουμε να πούμε ονόματο των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων κ και άλλα μέλη αναφέρθηκαν στο πρόβλημα που μας απασχολεί όλους με, το, με το, τα χρονικά περιθώρια, αν θέλετε. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες ανάμεσα στους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ευθύνη είτε πρόκειται για τροχαίο υλικό, είτε για ε, ενδείξεις, για σήματα κτλ. Ε, πρέπει να είναι όλη η γραμμή, αν θέλετε, των ευθυνών ε, σαφέστατη και θα πρέπει οι πόροι να κατανεμηθούν ανάλογα. Έτσι, γιατί αλλιώς αν δεν, υπάρχει το, ε, ε, δεν υπάρχουν επαρκείς ανθρώπινοι πόροι δεν θα μπορέσουμε να ε, πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Επίσης το έγκαιρο, αυτό το χρονικό περιθώριο αν θέλετε, είναι ζωτική σημασία για να πετύχουμε την πλήρη λειτουργικότητα. Τα θέματα τώρα για τις ευθύνες. Εάν μεταφέρουμε την, ε, τις αρμοδιότητες των, ή ε, στην ΕΡΑ, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για οτιδήποτε ε, αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι ήταν ελαττωματικό για τους κανόνες ασφάλειας, ποιος θα αναλάβει ευθύνη εάν υπάρχει ελαττωματικό υλικό ή εξοπλισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ε, διευκρινίσουμε πώς αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τα θέματα της ευθύνης ε, γενικότερα, αλλά και ποιος θα αναλάβει ουσιαστικά την ευθύνη, ποιος θα είναι υπεύθυνο για το υλικό. Ε, οι εθνικοί φορείς κυρίως έχουν κάνει την περισσότερη δουλειά, είτε μέσω υπεργολαβιών, είτε ε, ξεκαθαρίζοντας τις ευθύνες. Εξού και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αέρα η ΟΕΡΑ έχει τις, ε, τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους. Βέβαια δεν μπορεί να αποκτήσει τόσο, ε, τόσο ανθρώπινο ε, υλικό, έτσι ως δυναμικό συγγνώμη, για να αναλάβει όλες, όλους τους τις ευθύνες των εθνικών φορέων. Αυτό ούτως ή άλλως το θέλουμε και κάτι άλλο τώρα που το ξέχασα, αλλά τέλος πάντων σταματάω εδώ τώρα γιατί ξέχασα, ήθελα να κάνω και μια τρίτη παρατήρηση, την οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν την έχω κατά νου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κράμερ για τους ε, πρασίνους, τέσσερα λεπτά. Βεβαίως, θέλουμε να αναπτυχθεί ο ERA, να γίνει Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συντονισμού που να ε, εξασφαλίζει την ποιότητα και την τήρηση των προθεσμιών. Αυτό δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και τόσο μεγάλη ε, μεταβατική περίοδο, διότι πολλά έχουν γίνει ήδη ε, και ακούμε όμως πολλά που λένε ότι αν να προσέξουμε να διατηρηθούν οι εθνικές αρμοδιότητες. Εγώ λέω όσο πιο γρήγορα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο, το νέο επίπεδο, τόσο περισσότερο κέρδο θα είναι για όλου. Να μα εξηγήσετε γιατί χρειαζόμαστε τόσο μεγάλε μεταβατικέ περιόδου. Φυσικά δεν θέλουμε να καταργήσουμε τι εθνικέ αρχέ. Φυσικά έχουν ικανότητε που πρέπει να διατηρηθούν, αλλά κάποια τμήματα πρέπει να περάσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι απόλυτα σαφέ ότι οι εθνικέ αρχέ θα ε, ε, έχουν ε, λιγότερες αρμοδιότητες, άρα και λιγότερο προσωπικό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα Έχουμε το EATMS, είναι 6.000 χιλιόμετρα όπου δεν μπορεί να πάει καμία σιδηροδρομική μηχανή. Έχουμε δηλαδή επαναλάβει αυτό που υπήρχε σε κάθε κράτος. Γιατί κάθε εθνική αρχή ήθελε ε, να διατηρήσει τις ιδιαιτερότητές της, ε, ο κλάδος το έκανε γιατί αυτό δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αλλά αυτό είναι κατά της ευρωπαϊκής αποτελεσματικότητας. Για το EATMS είναι υπεύθυνη η ERA και κανένας άλλος. Να είναι απόλυτα σαφές αυτέ. Αυτοί πρέπει να ελέγξουν, πρέπει να δούνε αυτές οι εγκαταστάσεις ε, ε, δοκιμών και ελέγχου ε, πώς θα γίνουν συμβατές οι με τις δε. Πρέπει να είναι σαφές. Φυσικά η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ERA και εθνικών αρχών, εθνικών οργανισμών είναι βασικό θέμα, αλλά το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, δεν είναι παρθένο το έδαφος. Υπάρχει ήδη καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων. Αυτό έχει ήδη ελεγχθεί, έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, πρέπει απλώς να διευρυνθεί. Υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως, η χρηματοδότηση είναι θέμα. Πρέπει να πληρώνει κανείς τον οργανισμό αυτό ERA για τη χορήγηση πιστοποίησεων Δεν θα τα αναλάβει όλα βέβαια ε, ο οργανισμός αυτός, η ERA. Η Κομισιόν προτείνει 43 επιπλέον θέσεις. Επαρκούν. Αυτό πρέπει να το δούμε και κάτι αποτελεσματικό. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες ότι ε, ε, οι αποσπασμένοι πρέπει να έχουν έναν ανώτατο χρονικό όριο απόσπασης. Πρέπει λοιπόν να αλλάζουν κάθε 8 χρόνια έχουμε τους κανόνες και στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ότι πρέπει να αλλάζει κανείς θέση. Αν θέλουν να ενισχυθεί η ERA, βεβαίως ξέρουμε ότι αν αλλάζει ε, ε, συνεχώς το προσωπικό, τότε μειώνεται και η ποιότητα εργασίας. Παρακαλώ να βάλετε στην έκθεση ότι πρέπει να υπάρξει απόκληση από του ε, συνήθει κανόνε που προβλέπουν κινητικότητα του προσωπικού. Εάν δεν υπάρξει αυτή η απόκληση, θα έχουμε ε, καταστροφικές συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. άλλος ένας ομιλητής, παρακαλώ. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό για τον οργανισμό σιδηροδρόμων ε, στην ουσία αφορά και τα δύο προηγούμενα. Γι' αυτό παίρνω τον λόγο τώρα. Συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι. Υπάρχει ε, συνένεση για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό σημαίνει εναρμόνιση των κανόνων στο τεχνικό τομέα και για το υλικό. Αναμφισβήτητο. Αλλά πώς θα ενισχύσουμε λοιπόν τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού, του ευρωπαϊκού. Συμφωνώ με τους Ρικέ και Παρνιό που είπαν ότι υπάρχει μια διτή ανάγκη. Πρώτα απ' όλα επαρκής πόρη δεν μπορούμε να έχουμε φιλόδοξους στόχους για νέες αρμοδιότητες και ενίσχυση του ρόλου του οργανισμού αυτού, αν δεν έχει και τους αναγκαίους πόρους. Αυτή η αναντιστοιχία θα οδηγούσε σε αποτυχία, που θα είχε επιπτώσεις και στην ασφάλεια, αλλά γενικότερα τη φιλοδοξία που έχουμε για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το σύστημα πόρων σωστά και υπεύθυνα. Να εμείνουμε να υπάρξουν ε, πάνω από 43 θέσεις. Να είναι ένας οργανισμός που να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και καλύτερα. Μεταβατικές περίοδοι βεβαίως χρειάζονται. Χρειάζεται μια ε, διεθνής αρχή, αλλά αυτή η διεθνής αρχή δεν πρόκειται να καταργήσει ε, τις εθνικές αρχές ε, από τη μια μέρα στην άλλη. Και με τη μία αυτές οι αρχές, οι εθνικοί οργανισμοί υπάρχουν θα ξέρουν ότι θα υπάρχει ένας ανώτερος οργανισμός που θα ε, διαιτητεύει και θα καθορίζει ε, τις τεχνικές προδιαγραφές. Και τέλος, ε, προτείνεται ένας, ένα επίπεδο έφεσης. Αυτή η έννοια ταχείας αντιμετώπισης της Κομισιόν δεν νομίζω ότι είναι επαρκώς σαφής. Πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα σε πιο χρονικό διάστημα αυτός ο φορέας ενστάσεων θα πρέπει να δίνει τις γνωμοδοτήσεις του. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνέπεια για αυτήν την ενιαία πιστοποίηση για τα δρομολόγια και για τα εμπορεύματα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η φύση των ε, μεταφερομένων εμπορευμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να μιλήσω κι εγώ για τις τρεις εκθέσεις. Προέκυψε από τη συζήτηση ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως είπε ο κύριος Μπάχ, ο κύριος Κράμερ και ο κύριος Γκρός, απόλυτα ανόητο να σταματάνε στα σύνορα τα τρένα, ενώ είμαστε το 2013. Από το 69 ε, στείλαμε κάποιον στο φεγγάρι, αλλά τα τρένα μας ακόμη σταματάνε στα σύνορα. Α δούμε τι γίνεται στι αεροπορικέ μεταφορές. Αν είχαμε τέτοια συστήματα στις ε, εναέριες μεταφορές, τα αεροπλάνα Airbus δεν θα είχαν πετάξει ποτέ. Θα περίμεναν κάποια πιστοποίηση από όλα τα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θα υπήρχε ούτε Α320, ούτε Α380, ούτε κανένα άλλο αεροσκάφος. Δεν θα είχαν κατασκευαστεί. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσει αυτό ο σιδηροδρομικός τομέα. Συμφωνώ οι πόροι του ERA δεν είναι επαρκείς για να πούμε ότι θα τα αναλάβει όλα. Πρέπει να υπάρξει όμως μια ιεράρχηση. Καθορισμός ποιος έχει την τελευταία λέξη σε θέματα διαλειτουργικότητας και τεχνικών προδιαγραφών. Εδώ έχουν ρόλο και οι εθνικοί οργανισμοί να δίνουν κάποιες πιστοποιήσεις για κάποια θέματα που αφορούν μόνο το εσωτερικό τους δίκτυο. Τέλος. Όπως ε, κάθε φορά, υπενθυμίζω στην Επιτροπή μας, πριν πάρουν το λόγο, για τους ιδεοδρόμους μας, τους πολιτιστικούς, ε, που ορισμένες φορές σε πολλές χώρες ε, χρησιμοποιούν τα εθνικά δίκτυα. Τους ιστορικούς δηλαδή και πολιτιστικούς ιδιοδρόμους. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους οργανισμούς που θα έχουν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την πιστοποίηση και τους ελέγχους. Οπότε, Εύα, σύντομα παρακαλώ σύντομα. Άντε, να είμαι επίκη. Είπε για το 69, το 1969. Το 1969 τα τρένα από την Αυστρία στην Ιταλία μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα. Τώρα υπάρχουν κάποιες δυσχέρειε στι ορισμένε περιπτώσει, Πρόεδρος. Ναι, ναι. Μιλώντας για αυτού τους πολιτιστικούς και τουριστικούς ιδιοδρόμους, τελευταία φορά που είχαμε πλήρε διαλειτουργικό δίκτυο ήταν με τις ατμομηχανές αλλά και εγώ πρέπει να αποδεχθώ ότι δεν θα επιστρέψουμε στον ατμό. Βεβαίως, τώρα από τις Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο κάνεις πιο πολύ ώρα με το σιδηρόδρομο από ό,τι πριν από 50 χρόνια. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο κύριος Πακέ. Πρέπει να μιλήσουν και οι συγητές. Δύο λεπτά ο καθένας. Θα είμαι πάρα πολύ γενναιόδωρος και θα σας ε, δώσω 15 λεπτά, αλλά θα είμαι και αυστηρός. Επομένως, ο κύριος Πακέ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τη γενναιοδορία σας. Ελπίζω δεν θα, δεν είναι συνήθιο, mm. μην το, πάρετε σαν δεδομένο, μια φορά έγινε. Ωραία, το ξέρω κύριε Πρόεδρε, η, ε, η κατανόηση προς την Κομισιόν σας είναι, προς την Κομισιόν είναι γνωστή. Πολλά ακούστηκαν για το τέταρτο νομοθετικό πακέτο για τους σιδηροδρόμους, ε, ακούστηκαν πολλά για την λογική των προτάσεων. Δεν χρειάζεται να επανέλθω και να εξηγήσω γιατί υποβάλλουν αυτές τις προτάσεις. Οι συγητές, οι σκιώδεις συγητές ε, τα εξήγησαν πολύ καλύτερα από μένα. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για αυτές τις τρεις προτάσεις και ένα γενικό συμπέρασμα. Θα ξεκινήσω με, την, με τον ε, οργανισμό σιδηροδρόμου, τον ΕΡΑ, να απαντήσω σε κάποια σχόλια. Προφανώς ο οργανισμός αυτός οδηγός σιδηροδρόμου θα είναι το κεντρικό σώμα αν θέλετε, ο κεντρικός φορέας που θα ασχολείται με τα θέματα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας. Θα είναι ο ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο θα κινούνται όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει το παρόν πλαίσιο, να λάβουμε υπόψη μας ε, και το διαφορετικό δυναμικό των εθνικών συστημάτων, αλλά και τις διαφορετικές ε, διοικητικές ε, κουλτούρες και προσεγγίσεις που υπάρχουν. Εξετάσαμε, όπως και πολλά μέλη μας είπαν ότι θα έπρεπε να το κάνουμε, ε, τα θέματα της ασφάλειας ε, ε, στην, σε αεροπορικές μεταφορές, στην, στην αεροπορία. Είδαμε ότι όταν δημιουργήθηκε η η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ε, υπήρχαν ε, διάφορα θέματα που τέθησαν στο Κοινοβούλιο και συζητήθηκαν και για την ασφάλεια και τις σχέσεις ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Φορέα και τους Εθνικούς Φορείς. Ε, υπάρχει εδώ μία έννοια την οποία υποστηρίζουν πολλά μέλη και εδώ αλλά και στο Συμβούλιο ότι ο ΕΡΑ θα ε, συνεργαστεί στενά με τους εθνικούς φορείς. Οι εθνικοί φορείς ε, δεν θα εξαφανιστούν, θα παραμείνουν και θα ασχολούνται, αν θέλετε, με τις ιδιαιτερότητες των εθνικών ε, συστημάτων, αλλά και θα υποστηρίζουν το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, όπως είπε ο κύριος Ρικέ ε, και άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Ζήλερ, ε, διότι εμείς είχαμε προτείνει ούτως ή άλλως 43 άτομα να προσληφθούν ακόμα στον οργανισμό, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, διότι δεν είναι καλά επανδρομένο εάν πρέπει όλες τις αρμοδιότητες που θέλουμε να τις αναλάβει, θέλουμε και 200 άτομα να έχει προσωπικό, αλλά τέλος πάντων οι 43 πιστεύω ότι θα είναι επαρκής έτσι ώστε να ε, μπορεί να εκτελεί το έργο το οποίο έχουμε, του έχουμε αναθέσει μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας απόφασης πάντα. Επίσης να ε, δημιουργηθούν και οι απαραίτητες ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει η συνεργασία. Εφόσον υπάρξει αυτή η συνεργασία ή το θέμα ευθύνης όμως θα το έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Ελπίζω ότι η προσέγγιση αυτή θα καλύψει κάποιες από τις ανησυχίες που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στις μεταβατικές περιόδους που πολλά από τα μέλη υπογράμμισαν. Στην πρόταση της Κομισιό έχουμε ε, μία κλιμάκωση αν θέλετε του ρόλου της, του ΕΡΑ στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Εμείς θεωρήσαμε ότι ούτως το 2015 θα ε, τεθεί σε λειτουργία η πρότασή μας και μετά στα, επόμενα τέσσερα χρόνια θα κλιμακωθούν οι δραστηριότητες ε, του ΕΡΑ. Προφανώς δηλαδή θα υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία και θα υπάρχει και ο χρόνος για να προετοιμαστεί ο ΕΡΑ για να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες που τους αποδίδουμε. Όμως ο οργανισμός αυτός Ευρωπαϊκός Οργανισμός έχει φτάσει σε ένα ε, επίπεδο ορίμανσης, αν θέλετε, που μπορεί να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της. Εδώ και έξι χρόνια λειτουργεί ε, και η ποιότητα του προσωπικού της ε, και η ποιότητα της εργασίας όσον αφορά την ασφάλεια μας αποδεικνύει ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της κλιμακούμενης δραστηριότητάς της θα μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα για τον ΕΡΑ, τα θέματα της ε, ευθύνης, ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά κατά την άποψή μου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα ευθύνης που αναλαμβάνει το προσωπικό και ο ΕΡΑ, ε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο ρόλο ε, του, του ΕΡΑ ε, θα πρέπει να ενδυναμωθεί, να ε, διευκρινιστούν περαιτέρω τα θέματα των, της ευθύνης και αυτό θα το αναλάβει και η Ιρλανδική Προεδρία. Τώρα, στα θέματα της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας. Πιστεύω ότι εδώ η προσέγγιση είναι παρόμοια η πρόταση είναι να αποχωρήσουμε σταδιακά από τους εθνικούς κανόνες που συνυπάρχουν ε, με τους ε, ευρωπαϊκούς και να μιλάμε ε, για πιστοποιητικά που θα στηρίζονται σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι εθνικοί κανόνες, αυτοί που είναι κοινοποιημένοι, είναι διάφανείς και χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό, θα αποτελέσουν κομμάτι της διαδικασίας Όμω Όμως θα υπάρχει ένα ενιαίο πιστοποιητικό το οποίο θα χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Εδώ λαμβάνουμε υπόψη μας και την υπάρχουσα διαδικασία όπου η εθνικοί φορείς σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό ε, εξετάζουν τους εθνικούς κανόνες που είναι και μια κληρονομιά του παρελθόντος. Σε πολλές περιπτώσεις έχει υπάρξει μια τροποποίηση ε, των κανόνων. Επομένως, επαναλαμβάνω ένα ενιαίο πιστοποιητικό το οποίο θα χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για την ασφάλεια, να σας πω ότι και για την διαλειτουργικότητα και για την ασφάλεια και για την αναδιατύπωση στα θέματα ασφάλειας ε, συζητήσαμε ε, λεπτομερώς μέσα στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας και οι τρεις προτάσεις αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας και υπάρχει σαφής ε, κατανομή ευθυνών και ανάμεσα στους εθνικούς φορείς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, αλλά και ανάμεσα σε αυτές τις επιβλέπουσες αρχές, αλλά και στις ε, συνδρομικές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε ένα καλύτερο, ένα πιο ασφαλές πλαίσιο. Επίσης πιστεύουμε ότι με αυτή την προοδευτική μεταφορά των ευθυνών προς τη και των αρμοδίτων προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων θα αποδεσμευθούν ε, ε, άτομα ε, και πόροι από, την, ε, από τους εθνικούς φορείς που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με, με χαρτιά ε, και θα μπορέσουν να ασχοληθούν πλέον με πιο πρακτικά και τεχνικά θέματα ασφάλειας. Αυτά είναι βέβαια θέματα τα οποία θα συνεχίσουμε να συζητάμε, αλλά πιστεύουμε ότι το νέο πλαίσιο το οποίο δημιουργείται θα ενισχύει περισσότερο τα θέματα ασφάλειας μία, δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις τώρα ε, σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν ε, οι βουλευτές. Το ένα αφορά το διοικητικό άχθος και τον κίνδυνο που υπάρχει οι άδειε ή τα πιστοποιητικά να αμφισβητηθούν, αλλά και ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο καλύπτει η πρότασή μας ε, που είναι το ότι το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να ανανεωθεί εφόσον δεν ανανεώνεται το υλικό ή μια συνδρομική η εταιρεία δεν αποφασίσει να λειτουργήσει και σε μια άλλη χώρα. Επομένως, ε, η πρόταση τη Κομισιόν λέει ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν αμφισβητούνται εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή. Και η δεύτερη, το δεύτερο σχόλιο, διότι εδώ ε, μιλάμε για τις ε, συνδρομικές εταιρείες και για τροχαίο υλικό, μιλάμε για σταθερό υλικό και η ευθύνη σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν ε, είναι κεντρικό θέμα της πρότασής μας. Δεν είναι βέβαια πολύ απλά τα θέματα, οφείλω να ομολογήσω και ε, ε, πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο και θα παραμείνουν αντικείμενο στον, ε, της διαθεσμικής συνεργασίας. Εδώ ολοκληρώνω ευχαριστώντας σας και τα μέλη για την συνεργασία. Ο τεχνικός πυλώνας, αν θέλετε, του τετάρτου νομοθετικού προγράμματος για τους σιδηροδρόμους είναι... Ένα, είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη τεχνική πρόταση θα πρέπει οι συνομοθέτες να εξασφαλίσουν ότι στο τέλος της διαδικασίας θα έχουμε σαφείς κανόνες, θα έχουμε σαφή κατανομή των ευθυνών και των υποχρεώσεων και αν το κάνουμε αυτό, σε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε διδαχθεί τα μαθήματά μας από το πακέτο του 2008, το οποίο ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξο, οφείλω να ομολογήσω. Ευχαριστώ κύριε Πακέ οι συγητές για δύο λεπτά εάν έχουν να πούνε κάτι. Κυρία Ντεγκράντες. Α, όχι. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Η κυρία, για την κυρία Μπιλμπάου εννοούσα. Είμαι μικρόσωμη. Παρ' όλα αυτά υπάρχω. Είναι η δεύτερη φορά που δεν με βλέπετε κύριε Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα. Θα κρατήσω τα πιο θετικά, παρόλο που ως προς τη δική μου πρόταση δεν άκουσα συγκεκριμένη απάντηση. Όλοι συμφωνούν βέβαια ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού οργανισμού, ο οποίος θα προδιαγράφει τους κανόνες και θα μας οθήσει να έχουμε ένα σιδηροδρομικό κλάδο πιο ανταγωνιστικό και θα μπορούμε να προσφεύγουμε για να γίνει, όταν δεν γίνεται σωστά η μεταφορά και θα, πρέπει να, θα μπορούν να κατανέμονται σωστά οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες. Αυτό θα ωφελήσει τους χρήστες, θα έχουμε τη μονοαπευθυντική θηρίδα, Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον, ενδιαφέρουσα αυτή η δουλειά, έχω πλήρη εμπιστοσύνη, πιστεύω ότι θα κάνουμε το απαραίτητο βήμα και θα είμαστε παράδειγμα για τον Ευρωπαίο πολίτη που περιμένει τέτοιου είδους αποφάσεις να λαμβάνουμε εμείς. Ευχαριστώ ο κύριος Κράμερ παρακαλώ. Και εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ένα <clears throat> είναι σαφές, σε ένα συμφωνούμε, ότι θέλουμε αυτά τα τρία πράγματα, πάντα τα θέλαμε αλλά ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Ευτυχώς έχουμε την πύρα του παρελθόντος που δεν ήταν πάντα τόσο θετική, άρα θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Δύο ερωτήσεις κύριε Πακέ. Συμφωνείτε ότι η Κομισιόν θα έχει την τελευταία λέξη σε περιπτώσεις ε, δικογνωμιών. Εντάξει. Ξέρουμε που είναι οι αρμοδιότητες, αλλά εάν υπάρχουν δικογνωμίες, συγκρούσεις ε, και ε, εμπλακή και η ΕΡΑ θα έχει την Κομισιόν τελευταία λέξη και για την ανταλλαγή, ε, ανταλλαγή προσωπικού με την ΕΡΑ. Συμφωνείτε με αυτά που είπαμε. Ή εδώ υπάρχει μπλοκάρισμα. Δεν θα μπορούσα να υποθέσω κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα μια απάντηση. Ευχαριστώ Ρόμπερτ. Και εγώ ευχαριστώ Μπράιαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τον κύριο Πακέ για τα σχόλιά του. Πήρα ένα μήνυμα για την έκθεσή μου ε, για την ευθύνη για το, τη χρονική συγκυρία της μεταβατικής περίοδου. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν. Ο ΕΡΑ πρέπει να έχει περισσότερες ευθύνες, αλλά η προσέγγιση να είναι λογική. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Και στα 25 κράτη-μέλη όπου υπάρχουν σιδηρόδρομοι, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε κανείς να μην είναι σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι ήταν πριν, μετά τη μεταγραφή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Και θα πρέπει να αξιοποιούνται οι πόροι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι ανθρώπινοι πόροι. Η διοίκηση του ΕΡΑ ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει ε, με τη στελέχωσή της και με τους ανθρωπίνους πόρους. Και στη Βαλτική πριν από το δεύτερο ε, Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τρένα που συνέδεαν την ε, Ρήγα με άλλες πόλεις και τώρα δεν το έχουμε και το στρέφουμε προς τους Ιταλούς και Αυστριακούς συναδέλφους που ανέφεραν κάτι παρόμοιο προηγουμένως. Πράγματι, είχαμε εξαίσιες ατμομηχανές εκείνη την εποχή. Σας ευχαριστώ όλους λέει ο πρόεδρος. Δεν οδηγούσα εγώ τότε βέβαια. Δεν είμαι, καν, δεν είμαι ούτε καν εγώ τόσο μεγάλος ώστε να τα θυμάμαι. Ελπίζω όμως ότι οδήγησα σωστά αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ε, Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε για τα δικαιώματα των εν αέριων μεταφορών. Θα τα πούμε στις 3. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα, διευκολύνατε τη δική μου θέση και τη δική μου δουλειά. Θα τα πούμε πάλι στις 3.